Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, υποψήφιο επίτροπο για την ε, κλιματική δράση και την ενέργεια, κυρίον Μιγέλ Άρια Κανιέτα, σε αυτή τη δημόσια ακρόαση που διοργανώνεται από κοινό από την Επιτροπή για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Επιστηστική Ασφάλεια και την Επιτροπή Βιομηχανίας ε, Έρευνας και Ενέργειας. If you wait, I'm going to explain. Μισό λεπτό, θα σας εξηγήσω. Μισό λεπτό. Ο Μιγγέλ Άριας Κανιέτε είναι αυτή τη στιγμή μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν ε, βουλευτής από το 1986 με το 1999 και ήταν πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, Αλίας από το 1995 στο 1997 και πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης από το 1997 έως το 1999. Στην Ισπανία ήταν επανειλημμένα γερουσιαστής και βουλευτής, υπουργός γεωργίας από το 2000 στο 2004 και Υπουργό Γεωργίας ε, Επιστημισμού και Περιβάλλοντος από το 2011-2014. Στην τελευταία του ιδιότητα εκπροσώπησε την Ισπανία στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη συναντήση κορυφής των ΗΠΑ για την κλιματική αλλαγή στην Τόχα και την Βαρσοβία. Το χαρτοφυλάκιό του καλύπτει ε, ε, πολλά θέματα που είναι κεντρικά για την ε, λειτουργία των δύο επιτροπών μας. Όσον αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την οποία έχω την τιμή να, τις οποίες έχω την τιμή να προεδρεύω. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε δεσμευτεί για μια αποτελεσματική και φιλόδοξη πολιτική για το κλίμα για να μειώσουμε τις εκπομπές ε, αερίων θερμοκηπίου και για να έχουμε μια βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη. Ανάμεσα στις νέες προτεραιότητες, στις κύριες προτεραιότητες μας είναι να υπάρχει ουσιαστική ηγεσία της Ένωσης στις διεθνείς κλιματικές διαπραγματεύσεις εν ώψη της συνάντησης κορυφής στο Παρίσι του 2015. Η σημασία να υπάρχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την ενέργεια, για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 και η αναγκαιότητα να μεταρρυθμιστεί η αγορά ε, άνθρακα στην Ένωση και ιδιαίτερα το σύστημα ανταλλαγή ε, εκπομπών. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τι ε, κατευθύνε γραμμέ για την έγκριση τη Επιτροπή, το Κοινοβούλιο εκτιμά την ικανότητα των υποψηφίων επιτρόπων με βάση τις γενικές τους ικανότητες, τη δέσμευσή τους για τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και την προσωπική ανεξαρτησία. Επίσης, αποτιμά την γνώση τους του χαρτοφυλακίου και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Πριν την ε, ακρόαση, οι γραπτές απαντήσεις που μας έστειλε ο Επίτροπος έχουν διανεμηθεί. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου όλες οι άλλες ε, μεταφράσεις διανεμήθηκαν ε, στα μέλη σήμερα το πρωί. Πριν να σας παρουσιάσω τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η ακρόαση, θα δώσω το λόγο στον Σνάλφο Μπούζεκ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για την έρευνα, την, ένεργη, την βιομηχανία, την έρευνα και την τεχνολογία για τις αγωγικές του παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, συνάδελφε Λαβία. Συμπροεδρεύουμε αυτή τη συνεδρίαση και θέλω να καλωσορίσω τον υποψήφιο επίτροπο Μιγέλ Άρια Κανιέτε που είναι ευρωβουλευτής άρα είστε σας στο σπίτι σας και καλωσορίζω και όλου του συναδέλφου από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και την Επιτροπή Βιομηχανία συνεργαζόμεθα πολύ. Πρέπει να συνεργαστούμε και συνεργαζόμεθα. Ε, όταν ε, πρώτο εξελέγει Ευρωβουλευτή, ήμουν ε, μέλο και των δύο επιτροπών αυτών για πέντε χρόνια και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Σα καλωσορίζω λοιπόν όλους. Καλωσορίζω του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Κοινωνία, μη κυβερνητικών οργανώσεων εταιριών, κρατών μελών, και επειδή είναι δημόσια ακρόασή μας και μεταδίδεται στο διαδίκτυο από τον ιστότοπο του Κοινοβουλίου ζωντανά. Λοιπόν, η Επιτροπή μας είναι αρμόδια για την ενεργειακή πολιτική, που είναι πολύ σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου του μέλλοντος επιτρόπου. Έχουμε τρία ενδιαφέροντα θέματα. Ενέργεια, ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας και νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα τρία θέματα ε, είναι πολύ στενά συνδεδεμένα με τα θέματα του κλίματος. Είναι αρμοδιότητα της Ήτρα. καθώς και άλλα. Η εσωτερική αγορά ενέργειας, η ασφάλεια της ε, προμήθειας ενέργειας, η προώθηση της ε, διασύνδεσης ε, των δικτύων, προώθηση των διευρωπαϊκών δικτύων, έρευνα ιδίω στον τομέα της ενέργειας, ενεργειακή ένωση. Όλα αυτά είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ήτρε. Άρα μας ενδιαφέρει πολύ να ακούσουμε τον κύριο υποψήφιο επίτροπο για το πώς προτίθεται να επιτελέσει το έργο αυτό. Και τέλος, η ενεργειακή μας πολιτική βασίζεται στο λεγόμενο τρίγωνο ενέργειας. Ασφάλεια, λογικές τιμές, προσιτές τιμές και περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω δράσης για το κλίμα. Χρειαζόμαστε μια σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών των στόχων. Αυτή η ισορροπία θα είναι βασικό καθήκον του Επιτρόπου για την κλιματική δράση και την ενέργεια. Και υπάρχει μια νέα ευκαιρία για μια νέα αρμονία μεταξύ των μέσων και στόχων μας. Και τέλος, είναι ουσιώδες για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας με βιώσιμο τρόπο, αλλά επίσης για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ενεργειακές κρίσεις και για να σταματήσει η ενέργεια να αξιοποιείται ως μέσο πολιτικής πίεσης, ως όπλο. Πολλούς στόχους λοιπόν έχουμε ενώπιόν μας για την επόμενη πενταετία και θα συνεργαστούν οπωσδήποτε και οι δύο επιτροπές και αυτή η πρώτη ε, κοινή συνεδρίαση είναι μία απόδειξη της ε, θέλησής μας να συνεργαστούμε. Παρακαλώ κύριε Λαβία, σας δίνω και πάλι το λόγο. Έχει ζητηθεί διαδικαστικό. Με συγχωρείτε, αλλά πριν προχωρήσουμε στην ακρόαση, έχω ένα διαδικαστικό από πλευρά τη Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Τι τελευταίε ε, ώρε ώρες ο Επίτροπος κ. Κανιέτα άλλαξε τρει φορέ τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δημιουργεί σύγχυση για το εάν η νομική επιτροπή αποτίμησε σωστά εάν συμμορφούνται προ τι υποχρεώσει του. Γι' αυτό ζητώ επισήμω από εσά του δύο προέδρου των δύο επιτροπών ο κύριος Λαβία, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι διαδικαστικό. Είναι διαδικαστικό. Η κυρία Φαν Είναι πολύ σημαντικό. Καλώ τους δύο συμπροέδρους να έρθετε σε επαφή με τον πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων να βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Προέδρου έχει ικανοποιηθεί. Μπορούμε να κάνουμε την ακρόαση, να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, αλλά πριν αποτιμήσουμε τον υποψήφιο επίτροπο, θέλουμε γνωμοδότηση της νομικής επιτροπής για το ότι η αλλαγή του τις τελευταίες 72, συγγνώμη, ότι η δήλωσή του τις τελευταίες 72 ώρες έχει αλλάξει τρεις φορές. Αυτή είναι η αίτησή μου από πλευρά της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Πρόεδρος. Βεβαίως θα ελέγξουμε πριν την αποτίμηση. Και τώρα να σας εξηγήσουμε την ε, οργάνωση της ακρόασης. Ο υποψήφιος επίτροπος, ο υποψήφιος επίτροπος καλείται να κάνει μία εισαγωγική δήλωση. Στις προηγούμενες ε, ακροάσεις που έκανε η Επιτροπή Ήτρε είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε κι άλλε ακροάσεις όπως ξέρετε. Κάθε φορά η εισαγωγή ε, διαρκούσε 10 λεπτά. Για την Επιτροπή Περιβάλλον επίση ήταν 10 λεπτά. Αλλά θα σα δώσουμε λοιπόν 10 λεπτά. Κύριε υποψηφίε Επίτροπε, αν θέλετε να υπερβείτε τα 10 λεπτά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ισχύει και για τις άλλες ε, κοινέ ακροάσεις. Κύριε Επίτροπε, θα έχετε 5 λεπτά επίσης στο τέλος ε, της ακρόασης. Κατόπιν, μετά την ε, παρουσίαση, θα υποβληθούν 45 ερωτήσεις. Ε, θα ακολουθήσουμε ε, τη διαδικασία ping-pong. Ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά απάντηση. Χωρίς συμπληρωματικές ερωτήσεις, επερωτήσεις. Δεν θα χωρίσουμε τις ερωτήσεις ανατομής πολιτικής ή κατά πολιτική ομάδα. ο χρόνος ε, ομιλίας ε, θα κατανεμηθεί με τους ίδιους κανόνες με τους, οποίες, με τους οποίους ε, λειτουργούμε στην Ολομέλεια. Σας παρακαλώ να τηρήσετε όλοι το χρόνο ομιλίας σας. Μόνο 5 δευτερόλεπτα ανοχή θα υπάρχει. Και 10 δευτερόλεπτα για σας κύριε Επιτρόπε. Μετά από αυτήν την μικρή υπέρβαση θα κόβω το μικρόφωνο μου. Θα βλέπετε το χρόνο σας και τους αστερίσκους όταν τον υπερβείτε στην οθόνη μπροστά σας. Υπενθυμίζω ότι έχουμε ταυτόχρονη διερμηνία σε 23 γλώσσες. Μπορείτε λοιπόν να μιλήσετε και να ακούσετε τη γλώσσα σας. Α, σας παρακαλώ να μην μιλάτε υπερβολικά γρήγορα. Η συζήτηση μεταδίδεται ζωντανά από τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης όλα αυτά εγγράφονται, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και εκ των υστέρων. Να δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στον κύριο Κανιέτε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα ενώπιόν σας ως υποψήφιος ε, για να αποτελέσω μέλος του επιτελείου του πρώτου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξελέγει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, βρίσκομαι μπροστά σας ε, έχοντας περάσει 13 χρόνια στα έδρανα αυτά χρόνια που τα θεωρώ από τα καλύτερα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας και του πολιτικού μου βίου. Γνωρίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γνωρίζω ότι ανέκαθεν υπεράσπιζε το ευρωπαϊκό συμφέρον και τις ευρωπαϊκές αξίες. Τις οικουμενικές αξίες της δημοκρατίας, ελευθερίας, δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και ισότητας που είναι τα θεμέλια που έκαναν την Ευρωπαϊκή Ένωση από τι πιο ευημερούσε και ελεύθερε περιοχέ του πλανήτη. Είναι αξίε που μα ενώνουν ω Δημοκράτε και Ευρωπαίου και διαπότιζαν ανέκαθεν την πολιτική μου δράση και αυτό θα κάνω και στο μέλλον. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην αρχή τη ισότητα. Στην προεκλογική εκστρατεία που πέρασε, έκανα ένα ατυχέ σχόλιο που έθεσε ένα αμφιβόλο τη δέσμευσή μου υπέρ τη αξία τη ισότητα. Ήταν όντω ένα ατυχέ σχόλιο. Ζήτησα συγγνώμη και τότε και θα ήθελα και πάλι να ζητήσω συγγνώμη. Λυπάμαι. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σημαντικός ακρογωνιαίος λήθος ε, για να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη, πιο ευημερούσα και, πιο, ε, και μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω κάποιες πληροφορίες που κυκλοφόρησα τις τελευταίες μέρες. Δεν πραγματοποίησα καμία απολύτως αλλαγή στη δήλωση οικονομικών μου συμφερόντων ε, ως επίτροπος. Και όλες μου οι δραστηριότητες και οι επαγγελματικές και οι πολιτικές αντικατοπτρίζονται πιστά στη δήλωση αυτή. Σε ό,τι αφορά το πόθεν έσχεση του Ευρωβουλευτή, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι χθες έκανα την ενημέρωση της δήλωσης αυτής μετά από αλλαγή των περιστάσεων που αναφερόταν στην δήλωση αυτή. Ήθελα να συμπεριλάβω την ολοκλήρωση της πώληση των μετόχων των εταιριών Πετροκλής και του ΚΑΡ, όπως είχα προαναγγείλει. Ούτε εγώ, ούτε κανένα από το στενό οικογενειακό μου κύκλο δεν έχουμε κανένα δεσμό με τι επιχειρήσει αυτέ. Και μάλιστα από αυτή την άποψη πήγα πολύ πιο μακριά από τι απαιτήσει τη ισχύουσα νομοθεσία. Επίση, θα ήθελα να σα ενημερώσω για την παρέτησή μου από τη θέση του Προέδρου του Ιδρύματο ΦΑΕΣ μετά την, τον ορισμό, το διορισμό μου ω υποψηφίου επιτρόπου. Και επίση, συμπεριέλαβα στο, στη δήλωσή μου και το αξίωμα του Προέδρου τη Εθνική Εκλογική Επιτροπή του κομματό μου από το 2008 μέχρι το 2011. Αυτό το αξίωμα περιλαμβανόταν και στη δήλωση ε, συμφερόντων που υπέβαλα στην Επιτροπή και στο βιογραφικό που υπέβαλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα νευραλγικό σημείο της ε, δημοκρατικής ζωής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό είμαι υπέρ ενός σημαντικού διαλόγου μαζί του που θα αποτελέσει τη βάση οποιασδήποτε πρόταση θα υποβάλλω. Είμαι στη διάθεσή σας και πρόθυμος και εγώ και οι υπηρεσίες μου για να έρθω για διάλογο, εξηγήσει ε, και για να ακούσω τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο διάλογος μας βοήθησε να ξεπεράσουμε εθνικούς εγωισμούς υπέρ ενός κοινού σχεδίου αλληλεγγύης που αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μεγάλη αίσθηση ευθύνης αναλαμβάνω την ε, δέχομαι την πρόταση που μου έγινε για να λάβω την, το χαρτοφυλάκιο των κλιματικών αλλαγών και της ενέργειας. Οι δύο πολιτικές αυτές είναι πολύ σημαντικές και θα σημαδέψουν το πεπρωμένο των επερχόμενων γενεών. Έχω ακράδαντε πεπιθήσει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι θα εξασφαλίσουμε και την ανταγωνιστικότητά μα και θα δημιουργήσουμε και θέσει απασχόληση. Και φυσικά οι προσπάθειέ μα θα πρέπει να έχουν μια διαχρονικότητα και να είναι και αποτελεσματικέ και να έχουν και απτά αποτελέσματα. Πιστέψτε με, από την πολιτική μου πείρα ως υπουργό Περιβάλλοντος είχα πολύ αποφασιστική και ξεκάθαρη δράση ε, και στήριξα τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε στη, μάχη, αυτή. Συνεργάστηκα στενά με την Επίτροπο Κόνι Χέντεγκαρτ και θα ήθελα να ποτίσω φόρο τιμή στο έργο της και στους συνεργάτες της. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε θαραλέοι και φιλόδοξοι σε αυτές τις πολιτικές. Κατά τη γνώμη μου, η απόφαση να συνδεθούν οι κλιματικές αλλαγές και η ενέργεια είναι ένα σημαντικό μήνυμα που θέλει να δώσει για τις πολιτικές αυτές ο εκλεγμένος πρόεδρος Γιούγκερ. Θέλουμε μια φιλόδοξη πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές και μια ενεργειακή πολιτική με βιώσιμο χαρακτήρα. Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και μάλιστα είναι σημαντικό που και τα δύο αυτά θέματα εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιο του ίδιου επιτρόπου. Έτσι θα εξασφαλίσουμε συνοχή των πολιτικών και θα δημιουργήσουμε τις απαραίτητε συνέργειες για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και ισχυροί. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πλαίσιο για το 2030 για το κλίμα και την ενέργεια αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το θετικό χαρακτήρα αυτής της ολοκληρωμένης εστίαση προκλήσεις είναι πολλαπλές. Θα πρέπει με αποφασιστικό τρόπο να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να μειώσουμε την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, να δημιουργήσουμε ένα ενεργειακό σύστημα που θα εξασφαλίζει ενέργεια σε προσιτές τιμές για όλους τους καταναλωτές, να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού, να μειώσουμε την ε, εξάρτησή μας από τις εισαγωγές και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Και όλα αυτά θα τα επιτύχουμε αν συνενώσουμε τις προσπάθειά μας και δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο. Έχουμε τεράστιο δυναμικό. Η εντολή που ανέλαβα από τον εκλεγμένο πρόεδρο είναι σαφής. Είναι καταρχήν σημαντικό να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην Σύνοδο Κορυφής για το Περιβάλλον των Παρισίων του 2015. Γι' αυτό και θα ήθελα να επισημάνω το, τη σημασία να είναι, να είναι φιλόδοξο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου και σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για μια συλλογική ευθύνη που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε. Θα πρέπει να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστής ε, σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών αλλά και για βιώσιμες θέσεις ανάπτυξης. Θα ήθελα ο κόσμος να συνδέει, να κάνει το συνειρμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την Ευρώπη. Θέλουμε φυσικά και δίκτυα που θα είναι ε, σύγχρονα και θα μπορούν να εκμεταλλεύονται στο έπακρο το δυναμικό αυτών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλουμε να γίνει η Ευρώπη ε, η πιο αποδοτική ήπειρο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργεια. Ήταν σαφή ο πρόεδρο Γιούγκερ. 30% υποχρεωτική ε, ενεργειακή απόδοση για το 2030. Απαραίτητη προπόθεση. Και θα συνεργαστώ μαζί σα για να προωθήσουμε τι απαραίτητε πολιτικέ, ε, επιδιώκοντα φυσικά τη συνένεση. Όλα αυτά θα γίνουν λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία μιας στιβαρής ενεργειακής ένωσης και μιας διορατικής πολιτικής για τις κλιματικές αλλαγές θα αποτελέσουν σημεία κλειδιά για το μέλλον. Διανύουμε ταραγμένους καιρούς και η όλο και μεγαλύτερη αστάθεια στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δημιουργούν ε, προβλήματα και έχουν συγκεκριμένε συνέπειε. Γι' αυτό ύψιστη προτεραιότητά μου θα είναι η εξασφάλιση του ενεργειακού ε, ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο τον, οκτώ, το φθινόπωρο. Στι 26 Σεπτεμβρίου, ο Επίτροπο Έτιγκερ υπέβαλε πρόταση για συμφωνία μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία για να αποφευθούν προβλήματα στον ανεφοδιασμό σε φυσικό αέριο το φθινόπωρο. Εγώ πιστεύω στη διπλωματία και θεωρώ ότι θα πρέπει να πριτανεύσει η λογική για να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου όλοι θα βγούμε χαμένοι. Και προ αυτή την κατεύθυνση θα εργαστώ ε, άοκνα. Η τροτότητα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την ενεργειακή εξάρτηση είναι γνωστή. Γι' αυτό και η ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει να αποτελέσει πολιτική προτεραιότητα. Και από αυτή την άποψη, ω Επίτροπο Κλιματικών Αλλαγών και Ενέργεια, θα συμβάλλω υπό το συντονισμό τη Αντιπροέδρου για την, ε, για την Ενεργειακή Ένωση θα συμβάλλω στην δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενέργειας με μια φιλόδοξη πολιτική κλιματικών αλλαγών που θα στηρίζεται στους ακόλουθους πυλώνες. Καταρχήν, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση πέρα το 2020, κυρίως ε, στα, στα κτίρια, στις μεταφορές και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Επίσης θέλουμε μια ουσιαστική ενιαία αγορά της ενέργειας με ελεύθερη κυκλοφορία της. Γι' αυτό Χρειαζόμαστε διασυνδέσεις και δίκτυα απόλυτα ολοκληρωμένα μεταξύ τους και να θέσουμε ένα τέρμα στις ενεργειακές νησίδες, είτε είναι φυσικές είτε κανονιστικές, βάζοντας τους καταναλωτές στην καρδιά και το επίκεντρο των αποφάσεών μας. Θα πρέπει να μειώσουμε την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας νέες πηγές και διαδρομές εισαγωγής. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη διαπραγματευτική μας δύναμη και να χρησιμοποιήσουμε αμφίδρομες ροές ενέργειας. Γι' αυτό και το γρήγορο άνοιγμα του νοτίου διαδρόμου θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της ενεργειακής πολιτικής ε, υπέρ της διαφοροποίησης και της ενεργειακής ασφάλειας. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε την, την τεχνολογική ανάπτυξη και την ε, έρευνα σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε νέες τεχνολογίες με χαμηλή χρήση άνθρακα που θα είναι αποδοτικές ενεργειακά. Επίσης θα πρέπει να αυξήσουμε και την δική μας παραγωγή ενέργειας και να βελτιώσουμε το συντονισμό των εθνικών ενεργειακών πολιτικών προκειμένου ε, να είμαστε ενωμένοι απέναντι στις τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε και ένα νέο σύστημα κοινή ενεργειακής διακυβέρνησης για να εξασφαλίσουμε μια πραγματική κουλτούρα ενεργειακής συνεργασίας και σε περιφερειακό επίπεδο. Θα ήθελα να υλοποιήσουμε πλήρως το πλαίσιο του 2030, συνδυάζοντας όλους τους μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας. Και γι' αυτό θα σας υποβάλω για κάποιες ιδέες. Θα ήθελα να ενισχυθεί το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Προτεραιότητά μου είναι η έγκριση του αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς για να εξασφαλιστεί η διαρθρωτική σταθερότητα που χρειάζεται η αγορά του άνθρακα. Και επίση θέλω να ενισχυθεί αυτό το σύστημα για να εξασφαλίσουμε συμμόρφωση με τους κλιματικούς στόχους μετά το 2006 με αποδοτικό και ε, προσοδοφόρο τρόπο. Επίσης, μετά από ένα πολιτικό διάλογο μαζί σας, θα υποβάλω νομοθετική πρόταση προκειμένου η κατανομή των εκπομπών αερίου του θερμοκήπιου που δεν ανακαλύπτονται από το σύστημα εμπορία εκπομπών να κατανεμηθούν μεταξύ όλων των τομέων. Σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ, θα χρειαστούμε προσαρμογή και σταδιακή μετατροπή όλων των συστημάτων, προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητες ισορροπίε. Και τέλο, θέλουμε μια μετάβαση σε μια οικονομία που θα χρησιμοποιεί πολύ λιγότερο άνθρακα και που θα πρέπει να συνδυάζεται με την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη καθώ και την καινοτομία θα πρέπει ταυτόχρονα να καταπολεμήσουμε την ανεργία, ιδιαίτερα των νέων. Και από αυτή την άποψη ο πρόεδρος Γιούκερ θα υποβάλει μια πρόταση, ένα πακέτο για την απασχόληση με επενδύσεις που θα ανέρθουν σε 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε αυτά αποτελέσματα ώστε οι κλιματικές αλλαγές και η ενέργεια να αποτελέσουν προτεραιότητα και της μελλοντικής αυτής πρότασης και του πακέτου. Αυτό προποθέτει βέβαια συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και πολύ διάλογο. Η ενέργεια και το κλίμα δεν έχουν πολιτικά χρώματα, ούτε είναι σε αντιπαλότητα μεταξύ του. Θα πρέπει να κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια. Ούτε ένα άνθρωπο στον πλανήτη δεν θα μείνει στο απειρόβλητο των κλιματικών αλλαγών. Ούτε μια γωνιά στην Ευρώπη, ούτε ένα σπίτι, ούτε μια επιχείρηση δεν θα απαλλαγεί από τι συνέπειε και μάλιστα θα ζήσει τι συνέπειε και από ενεργειακή άποψη. Ε, δεν μπορούμε να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Το διακύβευμα είναι τεράστιο και για να ανταπεξέλθουμε από κοινού στη μείζων αυτή πρόκληση ζητώ την υποστήριξή σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να ξεκινήσουμε τώρα τον γύρο ερωτήσεων. Πινκ πόγκα. Ο κύριος Πίτα Λίζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε Επίτροπε. Ευχαριστώ για την ε, στεναρή δήλωσή σας. Η δήλωση πόθεν έσχες είναι σωστή και μπορώ να διευκρινίσω αγαπητοί φίλοι, κυρία Φαν Μπρέμπτ ε, την ερώτησή σας. Έχω ένα email από τον Γενικό μας Γραμματέα Κλάους Βέλε και τον ε, αρμόδιο Γενικό Διευθυντή που λένε ότι υπήρξε ένα λάθος στη διοίκηση του Κοινοβουλίου και γι' αυτό φαίνεται ε, τρεις φορές να υπάρχει αλλαγή. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα το οποίο λύθηκε, δεν έχει να κάνει με τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Επίσης, είχε την καλοσύνη να μην κατηγορήσει τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, να μιλήσω για την κλιματική αλλαγή, κύριε υποψήφια επίτροπε. Ε, δείξατε μεγάλη δέσμευση για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά ξέρετε ότι ορισμένοι ακόμη και εδώ θεωρούν ότι το πρόβλημα είναι υπερβολικό, ότι ορισμένοι υπερβάλλουν, ότι δεν υπάρχει ε, καθόλου ε, ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή. Πώς αντιδράτε σε αυτές τις δηλώσεις. Ευχαριστώ για την ερώτηση. νομίζω ότι από το 1988 όταν δημιουργήθηκε το πάνελ IPPC για την κλιματική αλλαγή έχει κάνει θαυμάσια δουλειά. Έχουν κάνει πέντε διαδοχικές ε, αποτιμήσεις. Ε, κάθε φορά καταδεικνύεται όλο και περισσότερο ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και οφείλεται σε ανθρωπογενείς παράγοντες. Αυτό είναι σαφές. Πάνω από 2.000 επιστήμονες εργάζονται στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Συνεχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει χρηματοδοτήσει πολλή έρευνα για τους τομείς αυτούς μέσω των προγραμμάτων πλαίσιο. Και τώρα έχουμε το Horizon 2020 που χρηματοδοτεί έρευνα για την κλιματική αλλαγή. Έχουν τεθεί λοιπόν οι αποδείξεις ενώπιόν μας. Οι τρεις ε, τελευταίες δεκαετίες είναι η μία θερμότερη από την άλλη. Από τότε που έχουμε στοιχεία για, την, ε, για, τα, για το κλίμα δεκαετία του 50. Οι ωκεανοί γίνονται πιο ζεστοί, οι πάγοι λιώνουν, τα ακραία φαινόμενα είναι όλο και πιο έντονα. Το βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Δεν μπορούμε λοιπόν να καθυστερήσουμε. Πρέπει να δράσουμε. Πρώτα απ' όλα να τονίσουμε ότι ισχύουν αυτές οι εκθέσεις των επιστημόνων και μετά να τις μετατρέψουμε σε πολιτική δράση. Να αξιοποιήσουμε αυτές τις εκτιμήσεις για να έχουμε φιλόδοξους στόχους στην ε, επικείμενη συνάντηση κορυφής στο Παρίσι. Και πρέπει επίσης να κάνουμε μια τεράστια επικοινωνιακή δουλειά έναντι της κοινή γνώμης, γιατί αυτοί που αντιδρούν και αρνούνται την ε, κλιματική αλλαγή είναι πολύ ισχυροί, έχουν πολλές δυνατότητε ενώ εμείς που ε, στηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει δράση, πολλές φορές είμαστε υπερβολικά επιφυλακτικοί. Θα κάνω λοιπόν πολλές ομιλίες τονίζοντας ότι ε, οφείλεται σε εμά η κλιματική αλλαγή και δεν είναι μόνο το διοξείδιο του άνθρακο, είναι επίση και το υδρογόνο, διάφορα οξύδια του υδρογόνου και το μεθάνιο. Και θα είμαι πολύ ενεργό προ αυτή την κατεύθυνση. Συγγνώμη, οξύδια του αζότου. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Φαν Μπρέντ. Ευχαριστώ. Κύριε Λίζα, έτσι καλλιώς θέλουμε να περιμένουμε την αξιολόγηση της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων. Δεν το χρειάζομαι το mail σας. Κύριε Υποψήφια Επίτροπη, για την ε, δήλωση σύγκρουση εφερόντων θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Πολύ πρόσφατα ανακοινώσατε ότι πουλήσατε τις μετοχή σας στην πετρολίφερα Ντούκαρ και την πετρολίγης Κανάρια. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν να σας κάνω και θέλω απάντηση με ναι ή όχι. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο γιο σα πριν από λίγε μέρες ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και στις δύο αυτές επιχειρήσεις, ότι ο γαμπρός σας σα αντικατέστησε στην Προεδρία και των δύο αυτών εταιριών και είναι αλήθεια ότι η δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη ε, μέτοχη της Πετροφιλέρα είναι εκείνοι που πήραν ε, μέρος ε, αυτών. Μπορείτε επίσης να μας διασφαλίσετε ότι θα τηρήσετε τις υποσχέσεις σας. Εσείς είπατε ότι ποτέ δεν θα ασχοληθώ με θέματα του χαρτοφυλακίου μου εφόσον συγκρούονται αυτά με συμφέροντα που έχουν να κάνουν με την οικογένειά μου. Κλείνει το μικρόφωνο της κυρίας Βαν Απάντηση. Θα σας τα διευκρινίσω όλα. Πρώτα απ' όλα, Με το που έμαθα ότι είμαι υποψήφιος επίτροπος για θέματα ενέργειας, φρόντισα να πουλήσω τις μετοχές μου και παρετήθηκε ο γιος μου. Δεν έχουν μετοχές ούτε θέσεις. Ούτε σε αυτήν την επιχείρηση, ούτε σε καμία άλλη επιχείρηση που να έχει σχέση με αυτήν. Σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Αλλά ας το δούμε κι αλλιώς. Γιατί δηλώνω ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και γιατί γιατί οι δύο αυτές επιχειρήσεις είναι δύο μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, 50 εργαζόμενους, είναι μικρές. Στα λογιστικά. Δεν κάνουν ούτε εξόριξη πετρελαίου, ούτε πουλούν καύσιμα, ούτε κάνουν επιθεωρήσεις εξορίξεων κλπ. Τίποτα από όλα αυτά. Πρόκειται για δύο μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχει λοιπόν σύγκρουση συμφερόντων. Αλλά προκειμένου να τα σχεδιάσω όλα καλά, πήγα ακόμα πιο μακριά. Πούλησα τις μετοχές μου και ο γιος μου παρετήθηκε. Ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο γιος μου έχουν θέσει σε επιχειρήσει αυτές. Ούτε σε καμιά άλλη επιχείρηση που να έχει σχέση με αυτές τις δύο επιχειρήσεις. Άρα δεν υπάρχει κανένα συμφέρον τη οικογένεια μου στις επιχειρήσει αυτέ. E Τώρα να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Κύριε Κανιέτα, 40% των στόχων μα για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2020 δεν είναι επαρκές. Και επειδή η σημασία του να έχουμε υποσχέσει ότι θα γίνουν ε, μειώσεις και από όλους μας τους εταίρους ε, στην ε, πορεία προς αυτήν την φάρσα του Παρισιού θεωρείται ότι θα πρέπει μετά την συνάντηση αυτή θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη, ένα άλλο καθορισμό των στόχων μετά τη συνάντηση στο Παρίσι. Πρώτον, θεωρώ ότι η πρόταση που είναι στο πακέτο για το 2030 είναι ισορροπημένη. 40% μείωση, 25% ανανεώσιμες και 30% ενεργειακή απόδοση. Που ο, Γιούνκερ είπε, είναι, ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι είναι το ελάχιστο απαραίτητο, το απόλυτο ελάχιστο και θέλει να είναι δεσμευτικό. Είναι λοιπόν ένα συνολικό και ισορροπημένο πακέτο. Θα χρειαστούν λοιπόν πολλές προσπάθειες από όλους τους τομείς, από όλους τους Ευρωπαίους για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Εάν εμείς φτάσουμε σε αυτή τη συνάντηση κορυφής και όλες οι άλλες οικονομίες του κόσμου, όλοι οι άλλοι μεγάλοι ε, όλες οι άλλες μεγάλες οικονομίες που εκπέμπουν συμφωνήσουν σε πιο φιλόδοξους στόχους Φυσικά δεν θα ήμουν κατά. Φυσικά η Επιτροπή δεν θα έχει αντίρρηση, δεν θα μπλοκάρει πιο φιλόδοξους στόχους. Αλλά αν γίνει κάτι τέτοιο, θα το δούμε. θα δούμε πώς θα συνδυαστεί με το στόχο του 40% για τα διεθνή πιστοποιητικά. Και επίσης ε, πρέπει να δούμε τι ήδη διεθνή πιστοποιητικά και τι ήδη διεθνείς πιστώσεις θα μπορούσαμε να έχουμε στη διεθνή αγορά και τι ποιότητα για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Γιατί δεν ήταν σαφής πάντα η κατάσταση με αυτούς τους καθαρούς μηχανισμούς ανάπτυξης. Ξέρω ότι θα έχω την υποστήριξή σας αν γίνω επίτροπος και θα εξετάσω πολύ προσεκτικά να δούμε τι ποιότητα θα έχουν αυτά τα διεθνή ε, πιστοποιητικά ή διεθνείς πιστώσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκερμπράντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, το χαρτοφυλάκιο, εδώ κάθομαι, για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, ίσω είναι το πιο σημαντικό από ολόκληρο το σώμα των επιτρόπων και πρέπει να ομολογήσω ότι δεν ήμουν υπέρ του να συγχωνευτούν τα δύο αυτά χαρτοφυλάκια. Αλλά Εφόσον η Επιτροπή πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και συνδυαστεί η ενέργεια με την κλιματική αλλαγή, ναι, μπορεί μάλιστα να επιτρέψει μεγάλη πρόοδο αν πάρουμε σοβαρά την πρόκληση αυτή. Οπότε η ερώτηση σήμερα είναι εξή. Εσεί, κύριε Κανιέτη, είσαστε ο κατάλληλο άνθρωπο για να αναλάβετε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Δεδομένου ότι τα συμφέροντα είναι και το μεγαλύτερο εμπόδιο στο να γίνουν οι αλλαγέ που πρέπει να γίνουν. Εσεί λοιπόν με το παρελθόν που έχετε, με τι σχέσει σα με τι πετρελαϊκέ εταιρείε, δεν φαίνεται να είσαστε ο σωστό άνθρωπο. Ένα τρόπο υπάρχει για να με πείσετε εμένα και την ομάδα μου ότι είσαστε ο κατάλληλο άνθρωπο. Αν μα δείξετε πόσο σοβαρά παίρνετε την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πείστε με λοιπόν για το προσωπικό σας αίσθημα για το ότι επήγει να γίνουν οι αλλαγές αυτές για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Απάντηση. Θα προσπαθήσω να σας πείσω. Αλλά πώς να σας πείσω. Κοιτάξτε. Ήμουνα υπουργό Περιβάλλοντος στην Ισπανία πριν τότε είχα τις μετοχές μου σε αυτές τις δύο μικρές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, πολεμούσα με την ε, Επίτροπο για το Περιβάλλον. Στο πλευρό της. Προκειμένου να προχωρήσουμε με το πακέτο 2030 για πολύ φιλόδοξους στόχους. Ήμουνα και μέρος της ομάδας Green Road στην Ισπανία. Δεν στήριζα το πετρέλαιο, αλλά τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, την, ε, ε, τον φοδιασμό ενέργειας. Έχω ήδη δουλέψει και πολεμήσει για να προστατεύσω τον πλανήτη από την κλιματική αλλαγή. Δουλεύουμε έτσι καλώς υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να έχουμε ομόφωνες συμφωνίες ουσιαστικά πρέπει 200 χώρες περίπου να συμφωνήσουν. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε χρέος στις επόμενες γενιές. Οι πολιτικοί δεν πρέπει να σκέφτονται βραχυπρόθεσμα, πρέπει να σκέφτονται μακροπρόθεσμα. Η κλιματική αλλαγή απαιτεί μακροχρόνιες, μόνιμες πολιτικές. Είμαι λοιπόν υπέρ αυτών και κατά το παρελθόν. Ποτέ δεν είχα συνδέσεις με το πετρέλαιο είχα ένα 2,5% σε αυτές τις εταιρείε. Όταν όμως είχα δημόσια ευθύνη και δημόσια καθήκοντα, δούλευα υπέρ των ελλακτικών πηγών ενέργειας, υπέρ της ασφάλειας εφοδιασμού. Αυτά κατά το παρελθόν και αυτά θα συνεχίσω να κάνω και στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Η συνάδελφος Ροντρίγες Ρούμπιο τώρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σα. Κύριε Αρίας Κανιέτα, πραγματικά έρχομαι σε δύσκολη θέση που θα πρέπει και εγώ να μιλήσω για την οικογένειά σας, αλλά το κάνω γιατί είναι απολύτως απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι δεν έχετε οικογενειακά συμφέροντα που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιό σας. Πολύ σπεσμένα ε, πουλήσατε τις μετοχές σας στις πετρελαϊκές εταιρείες Ντούκαρ και, και Αλλά ο κουνιάδο σα έχει άμεση σχέση με τι εταιρείε αυτέ. Δεν μα μιλήσατε προηγουμένω ε, για αυτόν τον άνθρωπο. Εκείνο ε, ε, συνεχίζει να έχει σημαντική θέση στι δύο αυτέ πετρελαϊκέ εταιρείε. Εγώ θα σας μιλήσω για ένα φίλο μου που είχε σπουδάσει τοπογράφος πριν την στεγαστική κρίση. Τελικά ασχολήθηκε με τους ηλιακούς θερμοσαρευτές αλλά η κυβέρνησή σα τότε καταπολέμησε τι ανανεώσιμες πηγές ενέργεια ε, και δώσατε έμφαση στις ε, βιομηχανίε εξόριξη. Και ε, ήσασταν κατά της αυτοκατανάλωσης. Ουσιαστικά επιβάλλετε κυρώσει έμεσα με την πολιτική σα Διακόπτει ο πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν, σε καμία περίπτωση δεν πώλησα εσπευσμένα τις μετοχές μου. Την Τετάρτη έμαθα από τον πρόεδρο Γιούνκερ ότι θα με προτείνει ε, για τη θέση του Επιτρόπου για το κλίμα και την ενέργεια και την ίδια στιγμή αποφάσισα να πουλήσω τις μετοχές μου για να εξασφαλίσω τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και ανεξαρτησία και να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία, καμία βιασύνη, μόνο διαφάνεια. η ακρόαση αυτή θα κρίνει αν είμαι κατάλληλο και επαρκή για επίτροπο. Οι επίτροποι είναι απολύτω ανεξάρτητοι από τι εθνικές πολιτικέ. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε υπόλογοι προ τι κυβερνήσει μα. Εμεί προασπίζουμε το κοινοτικό, το ενωσιακό συμφόρον. Τώρα, αν η Ισπανία υιοθετεί σφαρμένη πολιτική, εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το θέμα. Θέλω να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρωταγωνιστή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλω να τροποποιήσω τις, τα δίκτυα μεταφορών για να μπορέσουν και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να βρουν μια διέξοδο εκεί. Και θα σας δώσω και ένα αριθμό αν θέλετε. Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ισπανίας είναι 16,1% το 2013. Ο στόχος είναι 20% για το 2020. Η Ισπανία δηλαδή είναι από τις χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σωστό δρόμο γιατί έχει υψηλό στόχο για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα. Αλλά εμένα με ενδιαφέρουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές, η αναζήτηση των καλύτερων πολιτικών. Και επίσης ένα ενιαίο, ομοιόμορφο ευρωπαϊκό σύστημα στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να μην δημιουργηθεί στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και να μην τροχοπεδίσουμε την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτό θα το κάνουμε με τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος Έκχαλτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, πρώτα απ' όλα. Μπορείτε παρακαλώ να είσαστε σαφέστερος για το γαμπρό σας και τι σχέση έχει με τις διάφορες αυτές επιχειρήσεις. διότι δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Και έπειτα, δεύτερον, κάθε φορά σας παίρνει χρόνο για να αποκαλύπτετε νέα. Όταν, ας πούμε, για την πετρόλογης ε, Κανάρια το 2011 πήγαν χρήματα, εσείς ήσασταν πρόεδρος της εταιρείας αυτής και μόνο όταν αποκαλύφθηκε το 2014 είπατε ότι δεν το ξέρατε, δεν ξέρατε αυτή τη συμφωνία. Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρατε αυτή τη συμφωνία εφόσον ήσασταν πρόεδρος. Και το ίδιο και με τις μετοχές. Το ακούσαμε ότι μόλις ε, γίνατε υποψήφιος επίτροπος τις ε, πουλήσατε. Γιατί. Μόνο όταν ήσασταν ε, υπεύθυνο για την ενέργεια και το κλίμα. απάντηση. Όσο δεν είχα οριστεί υποψήφιος, δεν είχα κανένα λόγο να τις πουλήσω τις μετοχές αυτές. Είναι μια νόμιμη δραστηριότητα στην Ισπανία. Μόλις έμαθα ότι ήμουν υποψήφιος επίτροπος, ήμουν έτοιμος να τις πουλήσω, ξέροντας ότι δεν υπήρχε σύγκρουση συμφέροντος βασικά καθόλου. Αλλά προκειμένου να μην υπάρχει οποιαδήποτε πόνη πήγα και ακόμα πιο μακριά. Για να μην υπάρχει ακριβώς θέμα σύγκρουση συμφερόντων. Αποφάσισα, παρόλο που δεν ήμουν υποχρεωμένο, να τις πουλήσω και παρετήθηκα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν συμπληρώνει κανείς τη δήλωση αυτή, οικονομικών συμφερόντων και τον κώδικα διοντολογίας σας ρωτάνε ποια είναι τα συμφέροντά σας, τα δικά σας και της γυναίκας σας. Σας το λέω λοιπόν ότι ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο γιος μου, ούτε εγώ έχουμε κανένα συμφέρον σε καμία επιχείρηση. Είναι σαφές. Τώρα τι κάνουν οι άλλοι. Το θέμα είναι η στενή οικογένεια. Αυτό ρωτάνε. Και σας απάντησα γι' αυτό. Και το ξέρετε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Έδρασα μόλι έμαθα ότι ήμουν υποψήφιο επίτροπο. Όχι νωρίτερα γιατί νωρίτερα δεν μπορούσα. Έτσι και αλλιώ χρειάζονται τρει με πέντε μέρε στην Ισπανία για να πουλήσει μετοχέ. Δεν μπορεί να το κάνει αμέσω, γιατί πρόκειται για μια ιδιωτική περιορισμένη επιχείρηση. Με απόλυτη διαφάνεια λοιπόν προχώρησα και πήγα και ακόμα πιο μακριά από αυτό το οποίο μου ζητάτε. Και νομίζω ότι είμαι σαφής όταν λέω ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι η οικογένειά μου, η γυναίκα μου και ο γιος μου δεν εμπλέκονται στις επιχειρήσεις αυτές, ούτε και σε καμία άλλη επιχείρηση που έχει να κάνει με πετρέλαια. Ευχαριστούμε. Συνάδελφος Πεντιτσίνη τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Καλησπέρα κύριε Κανιέτε. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε για την οικογένειά σας. Εγώ θα σας μιλήσω για τη δική μου οικογένεια. Γιατί και εγώ και η οικογένειά μου και όλος ο λαός, όλοι οι συμπολίτες μου ζούμε σε μια περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί που χρησιμοποιεί τη υδρορογμάτωση για την εξόριση πετρελαίου εδώ και 20 περίπου χρόνια. Έχω λοιπόν εύλογους λόγους για να σας πω ότι στην πατρίδα μου έχουμε τεράστιο ποσοστό ανεργίας και νέων και παρόλα αυτά συνεχίζουμε να καταστρέφουμε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για να τις διαθέσουμε σε εξοριστικές βιομηχανίες. Για να μην μιλήσω για τα απόβλητα που δημιουργούν αυτές. Και επίσης έχουμε αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου που οφείλονται σε βαρέα μέταλλα ή σε εισπνοή τοξικών αερίων. Τι λοιπόν θα κάνετε για τη δημόσια υγεία, γιατί η ενθάρρυνση τέτοιων βιομηχανιών αποβαίνει μοιραία για την υγεία των πολιτών. Όπως ξέρετε, κύριε Βουλευτά, η συνθήκη εκχωρεί το αποκλειστικό δικαίωμα στα κράτη-μέλη να εκμεταλλεύονται και να διαχειρίζονται όπως επιθυμούν τον ορυκτό τους πλούτο και τις πηγές ενεργειάς τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέβαλε συστάσεις χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα προβλέποντας ότι σε περίπτωση που ληφθεί σχετική απόφαση, η εξόριξη θα πρέπει να γίνεται με βάση κάποιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το παρόν σύσταση έχει υποβάλει, χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα όμως έχει τεθεί σε ισχύ ένα δίκτυο, ένα επιστημονικό δίκτυο, που θα αναλύσει όλες τις εμπειρίες εξόρυξης και σχιστολιθικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα προγράμματα που ήδη εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη για να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές και οι συνέπειες για το περιβάλλον αυτής της μορφής εξόρυξης. Επίσης θα μπορούσα να προτείνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο για την εξόριξη σχιστολιθικού αερίου με βάση συγκεκριμένες ε, περιβαλλοντικές ε, προδιαγραφές και αυτό φυσικά θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Επίτροπο Περιβάλλοντος. Σας διαβεβαιώ ότι θα συγκεντρώσουμε και θα αναλύσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, ε, τις συνέπειες τους στα οικοσυστήματα, στους υδροφόρους ορίζοντες, τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες και με βάση αυτή την ανάλυση θα κρίνουμε αν είναι σκόπιμο να θεσπίσουμε δεσμευτικές διατάξεις για να ρυθμίσουμε το θέμα αυτό. Το θέμα δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί επαναλαμβάνω υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών για το θέμα αυτό, αλλά έχουμε και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαφυλάξει το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τα φυσικά ενδιατήματα, τους υδροφόρους ορίζοντες και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Πιλάρ gracias κύριε υποψήφια επίτροπε κύριε Αρία Κανιέτα. Ευχαριστώ για την σαφήνεια και την ε, αφοσίωση που ακούσαμε στην ομιλία σας για την κλιματική αλλαγή και για την ενέργεια. Σίγουρα θα επιμείνουν διάφοροι σε κάποια οικογενειακά ζητήματα σε όλη τη διάρκεια της συζήτηση γιατί εφόσον απεδείχθη ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων γιατί και ορισμένα πράξατε εσείς αλλά και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων τα έλεγξε, οπότε να περάσουμε στην ουσία. Εγώ θέλω να μιλήσω για θέματα ενεργειακής ανεξαρτησίας. Φυσικά η έλλειψή της οφείλεται σε έλλειψη και υποδομών που δημιουργεί αυτούς τους θύλακους και Επίσης μπορεί να βοηθήσει ανάπτυξη των εφείων δικτύων. Έχουμε πολλά ε, προγράμματα που έχουν υποβληθεί και δεν έχουμε επαρκές πιστώσεις. Τι θα αξιοποιήσετε εσείς για να, πιέσουμε να υπάρξει εξυγχρονισμό των δικτύων και να υπάρξει η αναγκαία διασύνδεση των δικτύων που είναι απαραίτητη. Προφανώς. Για να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια χρειάζονται διασυνδέσει στη Βαλτική, στην Ιβυρική Χερσόνησο, στην Ανατολική Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο, ενοποιημένο και ευφυέ δίκτυο που να το, μας επιτρέπει να αξιοποιούμε πλήρως ε, αυτές τις διασυνδέσεις. Η ελάχιστη δέσμευση που συμφωνήθηκε στην Βαρκελόνη το 2000 υπήρχε ένας ενδεικτικός στόχος 10% ε, ελάχιστο διασυνδέσεων. Ο στόχος αυτός ε, βεβαίως έχει εκπληρωθεί και με τα προγράμματα ενωσιακού συμφέροντος ε, θα προχωρήσουν για το φυσικό αέριο και την ενέργεια. Δυστυχώς υπάρχει μία εξαίρεση που μας ε, λυπεί ιδιαίτερα, είναι η Βυρική Χερσόνησο που είναι σαν νησί. Και πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε και σε αυτό. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή θέλει να ξεκινήσει διάλογος με τις ρυθμιστικές αρχές στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία για να ξεπεράσουμε αυτό το μπλοκάρισμα και υπάρχει ένα πρόγραμμα διασύνδεσης μέσω των Πυρηναίων που ήδη έχει ξεκινήσει ούτω ώστε να περάσουμε από τα 400 στα 800 ΜΒ αλλά ορισμένα άλλα είναι πολύ αργά. Για παράδειγμα να διασυνδεθεί η Ακουιτανία με τον δισκαϊκό κόλπο μέσω των Πυρηναίων. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια από την Επιτροπή γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα χρηματοδότηση. Πρέπει επίσης επειδή ε, οι δυνατότητες του διασυνδέοντας στην Ευρώπη δεν είναι αρκετές, να δούμε πού αλλού μπορούμε να βρούμε την αναγκαία χρηματοδότηση, για παράδειγμα από τα 300 δις του πακέτου Juncker, για να έχουμε συγκεκριμένες λύσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρότε. Τις τελευταίες εβδομάδες, κύριε Κανιέτε, η σχέση σας ε, και οι οικογενειακοί σας σχέσεις με την ενεργειακή βιομηχανία συζητήθηκαν πολύ και χθες ε, προσαρμόσατε και πάλι τη δήλωσή σας. αργά παρά ποτέ. Και για το backloading επίσης καθυστερήσατε, αλλά πολύ αργά και αυτό. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το σύστημα εκπομπών, το σύστημα ε, εμπορίας εκπομπών. Θεωρείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η δυνατότητα σταθεροποίησης της αγοράς ή θεωρείτε ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μετά το 2020 όταν ίσως να είναι πολύ αργά για αυτό το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών. Παρακαλώ, ε, είπατε ε, ήδη ορισμένα για την οικογένειά σας. Παρακαλώ οι στενείς συγκινήσει να μας πείτε πώς συνδέονται με αυτές τις επιχειρήσεις. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Γι' αυτό καλύτερα να απαντήσω στα αγγλικά. Δεν επαρκούν τα γερμανικά μου. Πρώτον, θεωρώ ότι η αγορά αυτή τη στιγμή είναι θαυμάσιο μέσο. Έχουμε ένα σύστημα τιμών για, το, για τα αέρια, άνθρακος, αλλά παρά τα προβλήματά το σύστημα αυτό λειτουργεί. Είναι επαρκές για να μας οδηγήσει σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων άνθρακο. Θέλω λοιπόν αυτό το σύστημα ETS να αναπτυχθεί περαιτέρω. Αλλά επίσης, με ρωτήσατε για το αποθεματικό για τη σταθεροποίηση τη αγορά, Νομίζω πως είναι ευφυές ε, όργανο, ευφυή μηχανισμό. Ε, αποφεύγει αυτά τα πολιτικά παιχνίδια με την τιμολόγηση της ενέργειας. Αν είναι υπερβολικά τα ποσά πάνω στο αποθεματικό, αν είναι ανεπαρκή, παίρνει από το αποθεματικό και μας επιτρέπει λοιπόν να λειτουργήσουμε. Με ρωτήσατε αν θα πρέπει να προχωρήσουμε ή όχι. Φοβάμαι. Θεωρώ ότι το backloading ήταν ε, κάτι που μπορεί να γίνει μόνο μια φορά. Και αυτά που έχουμε αφαιρέσει από την αγορά θα επανέλθουν. Άρα μπορεί να επηρεάσουν τις τιμές. Και αυτό θα ήταν ε, κακή εξέλιξη. Αν λοιπόν με υποστηρίξετε παρκώς εσείς εδώ, θα επιχειρήσω να πείσω το Συμβούλιο, ούτω ώστε το αποθηματικό για τη σταθεροποίηση της αγοράς να αρχίσει να εφαρμόζεται νωρίτερα. Γιατί αυτό θα αποτρέψει τις ε, στρεβλώσεις της αγοράς και ακόμη και τις διαταράξεις στην αγορά που μπορεί να προκαλέσει η επάνωδος του backloading. Αρκεί να έχουμε την πλήρη υποστήριξή σας για το μέτρο αυτό, γιατί όλα τα θέματα που σχετίζονται με το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι περίπλοκα. Χρειάζομαι λοιπόν την εκ των προτέρων στήριξή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιατσκέβιτς. Ευχαριστώ. Κύριε Κανιέται θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας υποβάλλετε τις ε, πρωτοβουλίες που σκοπεύετε να, να λάβετε για να ενισχύσετε την ε, ενεργειακή μας ανεξαρτησία ε, και ε, από προμηθευτές, διαδρόμους και διάφορα είδη και ποιες ενέργειες. Ποιες είναι οι προτάσεις που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει αυτή την ενεργειακή ανεξαρτησία. Επίσης, πώς θα στηρίξουμε τις τοπικές αρχές για να αξιοποιήσουν τις πηγές ενέργειάς τους. Τι συνέπεια θα έχει στην ευρωπαϊκή οικονομία και στην επαναβιομηχάνηση η μεταρρύθμιση που θα προταθεί για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ποιοι βιομηχανικοί τομείς θα υποστηριχθούν από το... και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα από το σύστημα εμπορίας εκπομπών όπως θα μεταρρυθμιστεί και ποιοι θα πληγούν από τις αλλαγές αυτές στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Ευχαριστώ. First of all, uh... Καταρχάς, πιστεύω ότι για να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές ανεφοδιασμού μας. Δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε από ένα και μόνο προμηθευτή για πετρέλαιο και ε, φυσικό αέριο. Και επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε τις διασυνδέσεις μας ανά την Ευρώπη. Θα πρέπει να αναπτύξουμε τον νότιο διάδρομο. Είναι σαφές ότι το South Stream δεν θα προχωρήσει αν προηγουμένως δεν ε, εφαρμόσουμε το σύνολο του κοινοτικού κεκτημένου. Αλλιώς θα μείνουμε εξαρτημένοι σε τρίτες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και φυσικά να αναπτύξουμε και κάποια προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης, θα πρέπει να βρούμε κονδύλια και από τα διαρθρωτικά ταμεία. Το 20% των διαρθρωτικών ταμείων αφιερώνεται στην καταπολέμηση των, ε, πολιτικών, κλιματικών αλλαγών και την ε, διόρθωση προβλημάτων στον ενεργειακό τομέα. Θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια. Επίσης, με ρωτήσατε πώς θα λειτουργήσει το μεταρρυθμισμένο σύστημα εμπορίας εκπομπών, το ETS, και πώς θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων της βιομηχανίας θα, έχουμε και το σύστημα των ε, δωρεάν αδειών για κάποια κρατημέλη. Των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών. Μερικά κράτη ήδη εφάρμοσαν αυτό το σύστημα και μάλιστα έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να δούμε τι αλλαγές θα επιφέρουμε ώστε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας ή και να τη βελτιώσουμε. Επίσης, θα πρέπει να ε, στηρίξουμε και τις χώρες που θέλουν να κρατήσουν κάποια ενεργειακά εργοστάσια, είτε ε, εφαρμόζοντας το παλιό σύστημα, είτε προβλέποντας συγκεκριμένες αλλαγές στο νέο σύστημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτερσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με δύο μεγάλες προκλήσεις σήμερα. Πρέπει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και πρέπει να βελτιώσει και την ενεργειακή μας ασφάλεια μέσω του ενεργειακού εφοδιασμού με τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και μειώνοντας την εξάρτησή μας από εισαγόμενα καύσιμα δεδομένης της δυνατότητας που υπάρχει για μεγαλύτερη παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενεργειών, αιωλική κλπ. Εσείς πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτές οι δυνατότητες που υπάρχουν για καθαρή βιώσιμη ενέργεια θα ληφθούν πλήρως υπόψη και θα χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς εσείς προσωπικά θα διασφαλίσετε μια πραγματική ενιαία ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη που είναι και το κλειδί για να λυθούν αυτές οι δύο μεγάλες προκλήσεις που έχει η Ευρώπη μπροστά της σήμερα. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα για να αναπτύξουμε τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Το μεγαλύτερο είναι ότι δεν έχουμε ακόμα μια εσωτερική αγορά που να λειτουργεί καλά. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί στην εσωτερική αγορά. Δεν υπάρχουν εφηδίκτια, για παράδειγμα, για να παίρνουμε την ε, ενέργεια κλπ. Συνεπώς, πρέπει να επενδύσουμε και προσπαθώ να αναπτύξω νέα νομοθεσία για μια ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Όταν γίνει αυτό θα έχουμε επαρκή δίκτυα. Θα έχουμε φορείς οι οποίοι συντονισμένα θα, δουν, θα δρουν και θα μπορέσουμε έτσι να αναπτύξουμε περισσότερο τις δυνατότητές μας. Βέβαια και σε περιφερειακό επίπεδο στη Βόρεια Ευρώπη, για παράδειγμα, πρέπει να στηρίξουμε προγράμματα όπως είναι η πρωτοβουλία για τα offshore δίκτυα και άλλα αντίστοιχα προγράμματα. Σε περιφερειακό επίπεδο προς το παρόν μέχρι να έχουμε ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά συστήματα. Άρα χρειάζεται η περιφερειακή ολοκλήρωση, διασυνοριακή συνεργασία και σιγά σιγά να προχωρήσουμε προς την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Πάντως το πρόβλημα με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας θα παραμείνει όσο δεν έχουμε προχωρήσει με τα δίκτυα. Άρα χρειαζόμαστε ευφύ δίκτυα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. Συγχρόνως πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λόμπες Περμέχο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Κανιέτε, θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας Είμαι γυναίκα, πολύ θα ήθελα να κάναμε αυτό το διάλογο μαζί, αλλά δυστυχώ δεν προλαβαίνουμε. Πάντω, η κυβέρνησή σα κατάργησε τι εναλλακτικέ ενέργειε στην ε, Ισπανία. Είπατε υπέρ του φράκινγκ, τη υδρορογμάτωση, υπέρ του λιγοπολίου του ηλεκτρισμού, αδιαφορώντα για τα εκατομμύρια ανθρώπου που υποφέρουν. Αυτό είναι το μοντέλο που θέλετε εσεί για την Ευρώπη. Πώ έρχεστε εδώ σήμερα και μα λέτε το αντίθετο από αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Έπειτα εσεί δεν έχετε καμία νομιμότητα για το χαρτοφυλάκι αυτό, γιατί υπάρχουν τα συμφέροντά σα. Κάθε μέρα αλλάζανε τα πράγματα. Χτε μάθαμε για την αναμειξή σα στην ε, εκλογική επιτροπή του Ισπανικού Λαϊκού κόμματο. Δεν μπορούσατε να μα το είχατε πει νωρίτερα. Οι πετρελαϊκέ εταιρείε. οι δημόσιε συμβάσει που έπαιρναν επιχειρήσει αυτέ, Πώ, πώς, με ποιο τρόπο. Όλα αυτά όμως περνάνε από μια ε, η επιχείρηση στην Ολλανδία. Διακόπτει το μικρόφωνο ο πρόεδρος. Απάντηση. Δεν κατάλαβα ποια ακριβώς είναι η ερώτησή σας. Θα προσπαθήσω όμως παρόλα αυτά να σας απαντήσω. Το είπα και νωρίτερα. Εδώ, αν αναλάβω τελικά το χαρτοφυλάκιο εγώ δεν θα υποστηρίξω καμία εθνική πολιτική, αλλά ευρωπαϊκέ πολιτικέ υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και διάρθρωση των αναλλακτικών πηγών ενέργεια. Να υπάρχει επίση όρις δράση στην Ευρώπη. Αυτό που έρχομαι εγώ να κάνω στην Ευρώπη είναι να ρυθμίσω την εσωτερική αγορά ώστε να υπάρξουν συστήματα στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και να αποφύγουμε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κάποιε χώρε όπω η Ισπανία, όχι με την κυβέρνηση όπου εγώ συμμετείχα, αλλά με προηγούμενε κυβερνήσει, οι οποίες δώσαν υπερβολικές επιδοτήσεις και έκαναν το παιχνίδι να μην μπορεί να παιχτεί τελικά. Και καταλήξαμε σε τεράστιο έλλειμμα. Γι' αυτό λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό που θα κάνουμε είναι να καθορίσουμε κανόνες για να υπάρχει ένα σύστημα στήριξης που να βασίζεται στην αγορά χωρίς να βαραίνει σε επιδοτήσεις από τις χώρες μέλη και να είναι ενιαίος ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτό αποτελεί εγγύηση για τον ανταγωνισμό όπως επίσης και με την ανάπτυξη των εφιών δικτύων. Σε αυτά θα αφιερωθώ ως Επίτροπος. Να δώσω πρόθεση σε μια φιλόδοξη πολιτική, ενεργειακή ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεσματικής ενεργειακής πολιτικής, θα στηρίξω μια πολιτική υπέρ των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, υπέρ της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών, ώστε η Ευρώπη να γίνει ανεξάρτητη, κάτι το οποίο τόσο πολύ χρειάζεται σήμερα από το φυσικό αέριο και να αποφύγει την απομόνωση που πλήττει κάποιες χώρες. Ευρωπαϊκές πολιτικές λοιπόν θα προσπαθήσω να βρω ό,τι καλύτερο ώστε να υποφεληθούν όλε οι χώρες μέλη, ακόμα και εκείνε που παλιότερα είχαν προβλήματα επειδή υιοθέτησαν λαθασμένε πολιτικές. Ευχαριστώ. Η κυρία Βιβασί. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, μία από τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η διαφάνεια και όταν εξετάσω τις σταδιοδρομία σας ως Υπουργός Περιβάλλοντος δώσατε άδειες εξόριξης στην εταιρεία Rapsol λίγο έξω από τις ακτές των Καναρίων. Πρώτον, πήρατε, 12, ε, πήρατε δεκάδες αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα από δημόσιες αρχές για να δούμε πώς δόθηκαν αυτές οι άδειες και τις απορρίψατε όλες. Δεύτερο λάθος. Γίνονται εξορίξεις στη Μεσόγειο γεωτρήσει στη Μεσόβιο, ενώ όλες οι βιομηχανίες, όλοι οι κλάδοι και οι δημόσιες αρχές ήταν κατά οι τουριστικές επιχειρήσει τα επιμελητήρια. Στα πλαίσια της αναθεώρησης των κανόνων για την αναθεώρηση της ασφάλειας των ε, πλατφορμών εξόριξη, τι ε, εμπιστοσύνη μπορούμε να σας έχουμε. Ευχαριστώ για την ερώτηση σας κυρία μου. Θα σας πω το εξής. Δεν ήμουν ο υπουργό της βιομηχανίας της χώρας μου δεν πήρα την απόφαση να δοθεί έγκριση για την εξερεύνηση για πετρέλαιο, γιατί αυτές τις δίνει το Υπουργείο Βιομηχανίας. Το μόνο που κάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η Ισπανία είναι κράτος δικαίου. Η αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται από εμπειρογνώμονε, όχι από πολιτικούς. Έχουμε διακεκριμένους εμπειρογνώμονε που κάνουν αυτές τις ε, μελέτες επιπτώσεων. Εάν είναι θετικές οι μελέτες, τότε χορηγούμε τις άδειε. Αν αρνητικές, τις απορρίπτουμε. Εγώ αρνήθηκα την δημιουργία του μεγαλύτερου διελιστηρίου στην Ισπανία γιατί η μελέτη επιπτώσεων ήταν αρνητική αλλά ποτέ δεν επιχείρησα να επηρεάσω μια τέτοια, έκτιμη, ε, μια τέτοια εκτίμηση άφησα τους αρμόδιους υπαλλήλους να πάρουν τις αποφάσεις, διότι αυτοί με βάση επιστημονικά κριτήρια πρέπει να αποφασίζουν. Οι αποφάσεις για περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται με πολιτικά κριτήρια, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Η οδηγία για την ε, εξερεύνηση πέραν των ακτών που ε, πρόσφατα τροποποιήθηκε. Έχουμε ένα σωστό μέσο που διασφαλίζει την ασφάλεια αν υπάρξουν ατυχήματα, έχει όλους τους προληπτικούς μηχανισμούς και συστήματα και θα δω πώς θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία και ενδεχομένως, αν χρειαστεί, θα ε, κάνουμε ακόμη πιο αυστηρή την πρόληψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήμουν υπουργό Περιβάλλοντος, άφησα τους εμπειρογνώμονές μου να εκφραστούν και ακολούθησα πάντα τις απόψεις τους. Δεν πήρα καμία πολιτική απόφαση για να στηρίξω ένα φίλο κτλ. Βασίστηκα στην καλύτερη επιστημονική αρρωγή που μπορούσα να έχω και ε, εμπιστεύομαι τους εμπειρογνώμονες, όπως τους εμπιστεύομαι και στα Ηνωμένα Έθνη. Κύριε Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος, έληξε ο χρόνος σας. Και τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Χέλμερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, υποψήφια Επίτροπε. Είμαι ο εκπρόσωπος για την ενέργεια Τη μεγαλύτερη βρετανική αντιπροσωπεία στο Κοινοβούλιο, εθνική αντιπροσωπείας. Ξέρουμε ότι δεν έχει υπάρξει 18 χρόνια καμία θέρμανση του πλανήτη, καμία αυτό τον αιώνα. Ξέρουμε επίσης ότι η τρομερή υπερβολική αφοσίωση στις ανανεώσιμες έχει δημιουργήσει πρόβλημα ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Και το ξέρουμε αυτό γιατί ο Επίτροπος Άιτιγκερ είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πια να πληρώσει μια μονομερή ενεργειακή πολιτική και ο προηγούμενος επίτροπος Τατζάνη είπε ότι οι τιμές ενέργειας δημιουργούν μακελιό για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Θα κάνετε κάτι για να λύσετε το πρόβλημα. Έχετε κανένα ε, σχέδιο για να αυξήσετε την ανταγωνιστικότητα. Θα διασώσετε τις οικονομίες μας από αυτήν την συμφορά για την ανταγωνιστικότητά μας που δημιουργήθηκε από τη μονομανία μας με τα πράσινα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Αλλά επιτρέψτε μου να διαφωνήσω όσον αφορά την θέρμανση. Δεν είναι θέμα άποψης, είναι θέμα στατιστικών. Κάθε τρεις ε, δεκαετίες αυξάνεται η θερμοκρασία. Είναι σαφές στοιχείο αυτό. Αυξάνεται η, η θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 0,3 και αν υπερβεί τους δύο βαθμούς ε, αύξηση θα έχουμε καταστροφικές συνέπειες. Πρέπει λοιπόν με βάση αυτήν την θεώρηση να δράσουμε. Βεβαίως έχουμε πρόβλημα με την ε, τιμή της ενέργειας, με τις τιμές της ενέργειας, γιατί δεν έχουμε επαρκής, ε, επαρκή αποθέματα φυσικού αερίου, εξαρτώμεθα από άλλους για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην τιμή της ενέργειας. Οπότε έχουμε πρόβλημα σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να αναπτύξουμε τις δικές μας πηγές ενέργειας. Γι' αυτό στηρίζουμε τις ανανεώσιμές μας, υποστηρίζουμε την ενεργειακή απόδοση και πρέπει επίσης να έχουμε περισσότερη διαφοροποίηση πηγών και να αυξήσουμε και τη δυνατότητα μεταποίησης ενέργειας. Γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε ως Ευρωπαίοι για να έχουμε περισσότερη αγοραστική δύναμη. Διότι αυτή τη στιγμή κάθε εταιρεία συνάπτει τις δικές της συμβάσεις. Ο σύνολο θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερες τιμές. Αν μπορούσαμε να έχουμε μια δυνατότητα από κοινού διαπραγμάτευσης για την αγορά ενέργειας. Θα κάνω ό,τι μπορώ να πείσω τους εμπλεκόμενους να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Συνολικά, τι πρέπει να κάνουμε. Να πούμε ότι δεσμευόμεθα να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, να το πούμε στο Παρίσι και να απαιτήσουμε όλες οι χώρες να αναλάβουν τις ίδιες ευθύνες για να έχουμε ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Η κυρία Γκόντιν. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επιτρόπε. Άκουσα κι εγώ και είμαι επιφυλακτική ως προς τη πιθανή σύγκρουση φερόντων που σας αφορά γιατί δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, όπως λέμε στη Γαλλία. Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις, ε, ε, στις υπεράκτηρες ε, παρόλο που τα περιβαλλοντικά τους αποτελέσματα είναι αφισβητήσιμα. Και από οικονομική άποψη δεν αναπτύσσονται όπως περιμέναμε. Σήμερα η αποτυχία ενός σχεδίου στη Βόρεια Θάλασσα δείχνει ότι η μεγάλη κλίμακος παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ανεμογεννήτριες είναι ανέφικτη. Ερωτώ λοιπόν, θα ζητήσετε ανάλυση οικολογικών και οικονομικών επιπτώσεων των ανεμογεννητριών, ιδιαίτερα των υπεράκτιων ανεμογεννητριών και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας θα ήθελα να πω ότι είναι καλό να συγκεντρώνουμε στοιχεία από όλα μας τα προγράμματα και να τα αναλύουμε για να δημιουργήσουμε μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Αλλά έχουμε πρόβλημα έλλειψης ενέργειας, ε, λοιπόν διασυνδέσεων και μεγάλα προβλήματα σε ορισμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα στη Βόρεια Θάλασσα, ε, δίκτυα υπεράκτια, προσπαθούν να συνδυάσουν διάφορες προσπάθειες και να αναμίξουν και τις περιφερειακές αρχές. Όχι μόνο για να έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το θέμα αυτό αφορά και το backup, το μηχανισμό backup, αλλά και το φυσικό αέριο. Και θέλουμε να λύσουμε το μείζον ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις όλων των ευρωπαϊκών σχεδίων και προγραμμάτων. Και αναλαμβάνω τη δέσμευση να ζητήσω μελέτες επιπτώσεων για όλα τα προγράμματα και τα σχέδια που θα προτείνω. Επιπτώσεων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών. Σας υπόσχομαι ότι για όλα τα σχέδια που θα υποβάλω θα ζητήσω προηγούμενη τέτοια μελέτη επιπτώσεων. Και επίσης ευρεία διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους. Χρειαζόμαστε τέτοια ευρεία διαβούλευση, ευρύ διάλογο και φυσικά μελέτες επιπτώσεων για να δούμε πώς επηρεάζουν συγκεκριμένα σχέδια την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ πάντως ότι όλες αυτές οι πτυχές θα πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώς. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρινς. Ευχαριστώ κύριε Προτινόμενο Επίτροπε. Το χαρτοφυλάκιο κλιματικές δράσεις και ενέργεια ε, εμπεριέχει έναν κίνδυνο γενή και ένα δίλημα. Έχουμε τη συλλογική ανάγκη μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και τη επιβράδυση των κλιματικών αλλαγών. Απ' την άλλη, έχουμε το συμφέρον των καταναλωτών και τη βιομηχανία για χαμηλό ενεργειακό κόστο, αύξηση τη ανταγωνιστικότητα και αύξηση των θέσεων απασχόληση. Ερωτώ λοιπόν, ποιο κατά τη γνώμη σα θα είναι ο ρόλο σα για να βρείτε αυτή την ισορροπία δεδομένη στις ανάγκες και τη ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή τη μείωση τη ενεργειακή μα εξάρτηση από εισαγόμενο αέριο και μάλιστα από τη Ρωσία. Πιστεύω ότι ίσως αυτό θα είναι το πιο δύσκολο δίλημα. Γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ενεργειακό ενεφοδιασμό για όλους τους Ευρωπαίους, αλλά σε λογικές τιμές, σε προσιτές τιμές. Και εδώ δεν αρκεί μία και μόνο δράση, αλλά πολλές δράσεις σε πολλά επίπεδα. Θέλουμε ενεργειακή απόδοση, γιατί με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης έχουμε και οικονομίες, αλλά και πιο εύκολα θα εξασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια. Λοιπόν, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, έχουμε την σχετική οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Βέβαια, οι διατάξεις θα ισχύσουν μετά από το 2020. Τι θα γίνει με, την, με το οικολογικό design και την ε, την επισήμανση, την, ενέργεια την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Επίση, με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια θέλουμε να έχουμε χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, φθηνότερες τιμέ. Οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ακόμη δεν έχουν αξιοποιήσει όλε τι νέε τεχνολογίε. Επίση, το θέμα τη δέσμευσης και αποθήκευση του άνθρακα. Είναι σημαντικό το CCS και φυσικά εξασφάλιση διασυνδέσεων και ο νότιος διάδρομος αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα. Θα πρέπει να έχουμε διασύνδεση και της Βαλτικής βέβαια. Και αυτή είναι απαραίτητη. Και θα δούμε τι θα γίνει με το συγχρονισμό των ηλεκτρικών δικτύων. Δαπανηρό εγχείρημα, αλλά το χρειαζόμαστε. Είναι απαράδεκτο τρεις φορές της Ευρωπαϊκής Ένωση να μην είναι συγχρονισμένες με το ευρωπαϊκό σύστημα. Όλες αυτές οι δράσεις θα γίνουν παράλληλα. Αλλά θα πρέπει και οι ανταγωνιστές μας, οι εταίροι μας να εστερνιστούν αυτές τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές για να μην έχουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεν είναι εύκολο πάντως να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ των χαμηλών ενεργειακών τιμών και τον, ε, του στόχου των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Μάρτιν Έντουαρτ. Κύριε Κανιέτα, ήσασταν υπουργό όταν η Ισπανική κυβέρνηση στις 30 Οκτωβρίου 2013 νομιμοποίησε την υδρορογμάτωση και ξεκίνησε τις ε, εξερευνήσεις για σχιστολιθικό αέριο. Και επίσης εγκρίνατε την πρώτη μεγάλη παράδοση καναδικών ε, σχιστολιθικών άμμων στην Ισπανία. Θεωρείτε λοιπόν ότι η υδρορογμάτωση είναι τόσο ακίνδυνη και είναι δυνατόν να την επιβάλλουμε στον πληθυσμό μας ενώ παντού στην Ευρώπη γίνονται διαδηλώσεις κατά της υδρορογμάτωσης, ε, γίνεται συλλογή υπογραφών και εδώ δεν επιτρέπεται από την κυβέρνηση υδρορογμάτωση. Πώς καταλήξατε σε άλλη άποψη στην Ισπανία και η διάσκεψη του Παρισιού που επίκειται. Μπορείτε να μας πείτε τι ύψος αερίων θερμοκηπίου που θα προκύψουν από την ε, ε, χρήση αυτών των μη συμβατικών ορυκτών καυσίμων. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η απόφαση να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες υδρορογμάτωσης και σχιστολιθικό αέριο είναι ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων με βάση τις συνθήκες. Άλλες κυβερνήσεις μπορούν να το επιτρέψουν και άλλες μπορούν να το απαγορεύσουν. Η Επιτροπή έκανε μία σύσταση. Εάν επιχειρήσουν να κάνουν υδρορωμάτωση... τι κατευθύντηρες γραμμές πρέπει να σεβαστούν όσοι ζητούν άδειε. Δεν ήμουν εγώ υπουργό που ενέκρινε την υδρορογμάτωση. Ως υπουργό, πριν τη σύσταση της Κομισιόν, ως υπουργό λοιπόν αποφάσισα ότι η υδρορογμάτωση θα υπόκειται στις πιο αυστηρές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή ήταν η απόφασή μου ότι η τρογμάτωση θα πρέπει να είναι αντικείμενο περιβαλλοντικών μελέτης επιπτώσεων με τα πιο αυστηρά, τα πιο σκληρά κριτήρια. Τώρα η Κομισιόν έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο για να δει τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Και με βάση ό,τι θα μάθουμε ουσιώδη επιστημονική, πρακτική επιστημονική γνώση, τότε αν αναγκαίο θα προτείνω την κατάλληλη νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό στη συνάντηση κορυφής στο Παρίσι. Τι θα κάνουμε. Θέλουμε μια δεσμευτική συμφωνία όλων των χωρών που έχουν αναλάβει δεσμεύσεις. Να δούμε σε ποιο κοινό έδαφο θα μπορούσαμε να καταλήξουμε. Εμείς είμαστε πρωτοπορία γιατί θα εγκρίνουμε τον Οκτώβριο ένα πολύ ουσιώδες πακέτο και το 40% είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος που προτείνουμε. Ευχαριστώ κύριε Βυσνιεύσκα. Σας ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιε, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ, ε, ε εκπέμπει λιγότερο από το 10% των παγκόσμιων ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μάλιστα θα μειώσουμε στο 4% το 2030. Τι πρόκειται να κάνετε στα πλαίσια του μελλοντικού ενεργειακού κλιματικού πακέτου μέχρι το 2030 προκειμένου να διασφαλίσουμε την επιβίωση των ενεργειοβόρων βιομηχανιών που είναι όμως απαραίτητες για την ε, επιβίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η γεωπολιτική κατάσταση και συγκεκριμένες ε, πρώτες ύλες. Μόνο έτσι ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τους στόχους αναλογικά με τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, πώς ε, θα, θα πείσουμε τους εταίρους μας όπως η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε που είναι οι, από τις χώρες που εκπέμπουν περισσότερες, περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου να μειώσουν αυτές τις εκπομπές. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε για να συμμορφωθούμε με τους στόχους μας για την ενέργεια και το περιβάλλον είναι να εφαρμόσουμε τους στόχους για το 2020. Γιατί έχουμε νομοθεσία, θα πρέπει να την εφαρμόσουμε με τους στόχους που έχουμε θεσπίσει. Γιατί πολλά, πολύ νερό θα περάσει από το βλάκι μέχρι το 2020. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους στόχους αυτούς στον διάμεσο διάστημα. Θα έχουμε την οδηγία για την ενίσχυση του ETS, του, του συστήματος εκπομπών και επίσης ε, τι θα κάνουμε στα οι εταίροι μας που εκπέμπουν ε, ε, αέρια του θερμοκηπίου να αναλάβουν και αυτοί και να υλοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Σε συνεργασία με την ύπατη εκπρόσωπο θα έχουμε διπλωματικές επαφές με τους εταίρους μας. Θα έχουμε συνεχείς τακτικές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, στο σημαντικό οικονομικό φόρουμ που είναι σημαντικό για τις ανεπτυγμένες χώρες που εκπέμπουν και πολλές εκπομπές. Ε, θα θέσουμε το θέμα και στο G7 και στο G20 για να ετοιμάσουμε τις δεσμεύσεις και φυσικά και οι διμερείς επαφές θα έχουμε με την Ινδία, την Κίνα που είναι σημαντικοί παγκόσμιοι παράγοντες αλλά και με τις αναπτυσσόμενες χώρες γιατί και αυτές θα πρέπει να αναλάβουν κάποιες δεσμεύσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής για το κλίμα των Παρισίων. Οπότε θα έχω επαφές και με λατινοαμερικανικές χώρες, με την ομάδα ΘΕΙΛΑΚ ώστε να υιοθετηθούν στο Παρίσι δεσμευτικοί στόχοι. Είναι σημαντικό να αναλάβουν όλες οι χώρες του κόσμου δεσμεύσεις για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστούμε, κυρία Μπέρνερ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, είμαι γυναίκα, αλλά θα σας κάνω μια περίπλοκη ερώτηση. Το να πετύχουμε μια παγκόσμια συμφωνία για την μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι ζωτική σημασία για να αποφύγουμε την κλιματική αλλαγή. Οι αιτίε όμως είναι πολύ ευρείε και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, έχει να κάνει με την ε, αποψήλωση, έχει να κάνει με άλλα θέματα όπως είναι η μετανάστευση κτλ. Τι λοιπόν στρατηγική θα ακολουθήσετε για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις αυτές και μην ξεχνάτε ότι όλε οι χώρε του κόσμου περιμένουν την Ευρώπη να έχει τον ηγητικό ρόλο. Λέτε ότι θέλετε η Ευρώπη να αποτελέσει, να αποκτήσει μάλλον ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση των κλιματικών αραγών. Ε, δεσμεύεστε και για δεσμευτικές ε, προτάσεις και μετά το 2020, ώστε όλοι να τηρήσουν τους κανόνες και να αποφεύγεται η αποψήλωση στις ε, υποανάπτυξη χώρες, για παράδειγμα. Και η λοτομία. Απάντηση. Πρώτα απ' όλα θα αναλάβω δράση σε όλους τους τομείς. Γιατί θα συνεργαστούμε και στο Λούλου και σε όλους εκείνους τους τομείς, γεωργία, μεταφορές, τα πάντα. Και αν θέλουμε μια φιλόδοξη πολιτική για την κλιματική αλλαγή, πρέπει να βοηθήσουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες προκειμένου να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Μια από τις, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στο Παρίσι θα είναι το οικονομικό πακέτο. Πώς θα πετύχουμε δηλαδή συμβασμούς με τις χώρες αυτές. Διότι εμείς έχουμε δεσμευτεί 100 εκατομμύρια δολάρια είναι το πακέτο. Και τώρα διάφορες χώρες ζητούν διαφορετικά πράγματα από το Πράσινο Ταμείο. Το οικονομικό πακέτο λοιπόν θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διασφαλίσει τη στήριξη των στόχων μας στο μέλλον. Με ρωτάτε επίσης πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της υλοτομίας και της αποψήλωσης. Κοιτάξτε, υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχει βιομάζα, και προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη χρήση της βιομάζας και στο σύστημα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη βιομάζα, αλλά να μην αυξηθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι τύποι βιομάζας που να είναι λιγότερο αποτελεσματικοί. Αυτό που μας ενδιαφέρει πάντως είναι να χρησιμοποιήσουμε τους λιγότερο επιθετικούς τρόπους ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον αλλά συγχρόνως να βοηθήσουμε τις υπονάπτυξη χώρες να πετύχουν τους στόχους που θέλουμε να θέσουμε και να έχουν τη στήριξή μας γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χωρίστη Αμπάουντς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Κανιέτε. Οι προτεραιότητες τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι σαφές. Αν μας αναφέρετε αυτές, ουσιαστικά αποφεύγετε τα πραγματικά θέματα. Δεν μιλάω σαν οικολόγος απαραίτητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω για την υδρορογμάτωση. Για να αποφασίσετε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία, επ' αυτού θα λάβετε υπόψη σας την άποψη των Ευρωπαίων πολιτών κατά της δροματωσής Δεύτερον, εκ μέρους Μπενέγα και της Αστούρ, που θυμούνται πολύ καλά πώς αντιμετωπίσατε εσείς την καταστροφή του Πρεστίζ. Πώς θα φροντίσετε να πιέσετε την Ισπανική κυβέρνηση για να αποφύγει τη χρήση υδροκιανίου στις διάφορες διαδικασίες παραγωγής. Απάντηση. Το Ισπανικό κράτος πρέπει να τηρήσει όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές όπως και οι υπόλοιπε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικιά μου υποχρέωση ως Επίτροπος είναι ακριβώς να φροντίζω να τηρούνται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρώτο λοιπόν ήταν αυτό. Δεύτερον, επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο και στο Πρεστής, το ατύχημα του Πρεστή. Είπατε ότι ήταν καταστροφική αντιμετώπιση μου. Τότε ήμουν υπουργό Αλία. Και τι έκανα, έκλεισα τον χώρο που ψαρεύαμε εκεί στην Ισπανία, ώστε ακριβώς να προστατεύσω την υγεία των ε, πολιτών. Για μένα αυτό ήταν το πρώτο, η υγεία των πολιτών. Και στη συνέχεια βοήθεια προς τους αλείς, ώστε οι αλείς να μην υποφέρουν από την καταστροφή αυτή και να μπορούν από την αρχή μέχρι το τέλος ε, να αποφύγουν τη ζημιά στα διάφορα ληφτικά πεδία. Σας καλώ λοιπόν, όποιος θέλει, ας πάει στην Ισπανία, στη Βόρεια Ισπανία, και δείτε πόσο καθαρές είναι οι ακτές εκεί. Αυτό έκανα τότε για το Πρεστής, καθάρισα και τις ακτές. Και όσον αφορά τώρα την υδρορογμάτωση. Κάθε χώρα μέλος είναι κυρίαρχη να πάρει τις αποφάσεις της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε υποχρεώνει τις χώρες μέλη να αναπτύξουν την τεχνολογία υδρορογμάτωσης, ούτε τους υποχρεώνει ούτε τους απαγορεύει. Απλώς πρέπει να τηρούν τους κανόνες. Αν αποφασίσουν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν την τεχνική υδρορογμάτωση, είναι υποχρεωμένε οι χώρες να έχουν την κατάλληλη τεχνολογία. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθεί να έχει όλα τα επιστημονικά στοιχεία που υπάρχουν, να έχει πραγματογνωμοσύνη και από την Ευρώπη αλλά και εκτός Ευρώπης, ώστε να φροντίσει να έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές για την υδρορογμάτωση σε συνεργασία με εσά και με το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα κάνει προτάσεις έχοντας συζητήσει με όλα τα διαφερόμενα μέρη και εσείς εκπροσωπείτε τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μαραγάλ, κύριε Αρίς Μιλήσατε για σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχή σας ε, σε εταιρείε ε, πετρελαϊκές, αλλά όχι για κάτι άλλο βαθύτερο. Αυτά που κάνατε σε φορολογικούς παραδείσους, ίσως να είναι νόμιμα αυτά, αλλά είναι απαράδεκτα από πλευράς ευρωπαϊκής ηθικής. Θεωρώ ότι είναι ασύμβατο να αναλάβετε τις ε, αρμοδιότητες που προτείνετε να αναλάβετε με αυτά που έχετε κάνει στο παρελθόν. Σέβομαι τις απόψεις σας. Δεν συμφωνώ με τον νόμο για τι ακτές ή για τον Εύρο που κάνατε. Όλα αυτά από πλευράς περιβάλλοντος ε, δεν είναι ε, σωστά. Και νομίζω ότι αυτά που κάνετε ως επιχειρηματίας είναι γνωστά. Σας ερωτώ, θα ε, συνεχίσετε εσείς η οικογένειά σας να έχετε οικονομικά ενδιαφέροντες επιχειρήσεις στις Αντίλες ή τον Παναμά και θεωρείτε ναι ή όχι ότι θα ήταν σκόπιμο να παρετηθείτε, γιατί έτσι πιστεύω ότι θα έπρεπε να κάνετε. Λόγω αυτών των πληροφοριών που λάβαμε. Θα σας απαντήσω με απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο. Εγώ ποτέ δεν είχα οικονομικές δραστηριότητες σε εταιρείε που να είναι σε φορολογικούς παραδείσους. Ούτε έχω ε, οικονομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες που να είναι σκοτεινές. Όλα όσα έχω κάνει τα έχω δηλώσει πάντα στις ισπανικές φορολογικές αρχές. Όλες μου, όλα μου τα οικονομικά συμφέροντα είναι όλα δηλωμένα στην εφορία και είμαι περήφανος γι' αυτό. Δεν έχω μετοχές σε καμία εταιρεία στο εξωτερικό. Είχα κάποιες μετοχές και τις ε, πώλησα διότι ήθελα να είμαι σε κατάσταση απόλυτης διαφάνειας. Και Νομίζω ότι κι αν ήξερε ο πρόεδρος Γιούνκερ ότι είχα ακόμη αυτές τις ε, ε, μετοχές θα με είχε προτείνει. Εγώ τις είχα και τώρα τις πούλησα. Δεν έκρυψα ποτέ τίποτα. Και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι έχω απόλυτα ήσυχη, απόλυτα ήσυχη τη συνείδησή μου γιατί πάντα πλήρωνα τους φόρους μου ως πολίτης και είμαι πολύ ικανοποιημένος και πολύ ήσυχος γιατί πάντα το έπραξα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Ταμπουράνο. Κύριε Κανιέτα, μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ασχοληθεί στην ουσία με τους ε, καταναλωτές που είναι πολύ σημαντική στον τομέα της ενέργειας και για το τι εκπομπές θα έχουμε. Σύμφωνα με μελέτες του ΟΣΑ καταλάβαμε ήδη το 2008 ότι 80% των αποφάσεων για την ενέργεια από τους καταναλωτές λαμβάνονται από τις γυναίκες. Οι γυναίκες που είναι εκείνες που επίσης χρησιμοποιούν περισσότερο ε, τις δημόσιες συγκοινωνίες. Θα σταματήσετε λοιπόν τις διακρίσεις ε, τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες. Θα διαμορφώσετε μια πολιτική στον τομέα της ενέργειας που να λαμβάνει υπόψη τις επιλογές των γυναικών. Είστε διατεθειμένος να υιοθετήσετε μία προσέγγιση ίσης αντιμετώπισης έναντι των ε, γυναικών, για παράδειγμα, επιτρόπων. Έναντι όλων των γυναικών που θα συζητήσετε, με τις οποίες, για παράδειγμα, θα συζητήσετε στα πλαίσια των ε, ε, επαφών σας με μη κυβερνικές οργανώσεις. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι θεμελιώδης πυλώνας για μια δημιουργία, για μια Ευρώπη απόλυτα καλύτερη χωρίς αποκλεισμούς. Πιστεύω απόλυτα στην ισότητα ανδρών και γυναικών και από τότε που έχω αρμόδι... υπεύθυνες θέσεις στην πολιτική, πολλοί Ισπανοί ευρωβουλευτέ το ξέρουν, πάντα ε, έδωσα στις γυναίκες θέσεις ε, μεγάλη υπευθυνότητα. Της μέγιστης ε, υπευθυνότητα η κυρία Φράγα για παράδειγμα, τη έδωσα τη θέση για την αλληλεία, την πιο σημαντική για την γεωργία και η υπηρεσία για την κλιματική αλλαγή έχει επικεφαλής μια γυναίκα και η υπηρεσία για τις μελέτες περιβαλλοντικών πτώσεων έχουν επικεφαλής γυναίκα. Έχω πλήρη συνείδηση το πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να λαμβάνουν θέσεις λήψη αποφάσεων και πάντα το έκανα αυτό σε όλη μου την πολιτική σταδιοδρομία και μπορείτε να το ελέγξετε Τούτο λεφθέντων. Έχω διαβάσει χθε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ξέρω ότι έχει επίπτωση η κλιματική αλλαγή στις γυναίκες. Ε, αναφέρθηκαν πολλά. Και επίσης αναφέρθηκε ότι πρέπει να είναι γυναίκες στις σημαντικές θέσεις όταν θα λαμβάνονται αποφάσεις για την κλιματική αλλαγή. Διότι ακριβώς ε, όταν μιλούσαμε για την έκθεση για τις επιπτώσεις ε, της κλιματικής αλλαγής στην οικονομία της Αφρικής είδαμε τι επιπτώσεις έχει στις γυναίκες, άρα οι γυναίκες πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Καταλαβαίνω ότι σας ενδιαφέρουν οι ε, απόψεις των γυναικών για τη διαμόρφωση των αποφάσεων. Και στο ιδιαίτερο γραφείο μου φυσικά θα υπάρχουν ε, ίσως αριθμός ανδρών και γυναικών και επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου μου θα είναι γυναίκα και θα επιδιώξω η ισότητα των δύο φίλων να είναι πραγματικότητα και στις γενικές διευθύνσεις που θα υπάγονται σε μένα. Και ε, αν ε, με τιμήσετε θα φροντίσω να είναι γυναίκα ή επαναλαμβάνω η επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου μου. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπάλτσο. nukleáris erőművek megítélése környezetvédelmi szempont. Όταν πρόκειται για θέματα πυρηνικής ενέργειας, τότε υπάρχουν ε, πολύ διαφορετικές απόψεις. Η πλειονότητα των ε, περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι κατά των πυρηνικών. Αλλά σημαντικοί Αμερικανοί ερευνητές κατέδειξαν ότι για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, τη θέρμανση του πλανήτη, ο, η παραγωγή ενέργειας από πυρηνικές πηγές είναι πολύ θετική. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι δεν παράγει ε, εκπομπές. Είναι καθαρή. Ε, οπότε ρεαλιστικά ε, μέσω πρόθεσμα δεν μπορούμε να ξεφύγουμε την ε, πυρηνική ενέργεια διότι ε, το χαρτοφυλάκιό σας ε, δεν αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ενεργειακή πολιτική. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα ποιες είναι απόψεις για την πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ, όπως έχω πει πολλές φορές μέχρι τώρα η απόφαση για την πηγή ενέργειας που θα αναπτύξει κάθε χώρα είναι θέμα της κάθε χώρας. Δεν είναι θέμα ότι ένας επίτροπος είναι περισσότερο υπέρ μιας ή άλλης πηγής ενέργειας. Ο επίτροπος έχει ως καθήκον να ρυθμίσει την παραγωγή αυτή. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει υπέρ μιας ενέργειας που είναι καθαρή, έτσι όπως η πυρηνική, που έχει βέβαια το πρόβλημα των αποβλήτων, και γι' αυτό και εμείς έχουμε τις οδηγίες για τα πυρηνικά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διασφαλίσει το ανώτατο επίπεδο προστασίας. Και αυτό ακριβώς είναι που έχουμε κάνει με τις οδηγίες για την πυρηνική ασφάλεια και με τις οδηγίες μας για τα απόβλητα. Δουλεύουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, συνεργαζόμαστε με την Euratom και διασφαλίζουμε ότι αν υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να αναπτύξουν την πυρηνική ενέργεια, μπορούν να το κάνουν εφόσον διασφαλίζουν προστασία. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε φορά που υπάρχουν προγράμματα από τις χώρες μέλη τα μελετούν και κοιτούν ποιοι μπορεί να είναι οι περιορισμοί σε αυτά. Από εκεί και πέρα οι χώρες μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια πηγή ενέργειας θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες ε, στοιχηματίζουν στην πυρηνική ενέργεια, άλλες τις καταργούν όπως η Γερμανία και το Βέλγιο και άλλες θέλουν να φτιάξουν νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες, νέα, νέες τέτοιες μονάδες όπως η Ουγγαρία για παράδειγμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε οι διαδικασίες ε, ε, κατάργησης των ε, πυρηνικών μονάδων γίνονται βάσει συγκεκριμένων κανόνων και ότι τα απόβλητα πηγαίνουν στους χώρους που προβλέπεται για αυτά και όταν υπάρχουν νέες πυρηνικές μονάδες αυτές να χτίζονται βάσει των πιο σύγχρονων προδιαγραφών για να διασφαλίσουμε προστασία από την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη. Τώρα θα περάσω την Προεδρία στο συνάδελφο Μπούζεκ, ο οποίο θα αναλάβει το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας, της ακρόασης αυτής. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ Τζοβάνι. Έχουμε περάσει από τη μία πολιτική ομάδα στην άλλη. Περνάμε στον επόμενο γύρο. Ο συνάδελφος Ιβο Μπέλετ είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, εδώ είμαι μπροστά σας. Εκτιμώ πάρα πολύ την δέσμευση που αναλαμβάνεται απαντός ε, στον κύριο Κρότε όσον αφορά την μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ξέρετε ότι είμαστε σύμμαχοι στον ε, τομέα αυτό και ξέρετε πόσο πολύ μας ενδιαφέρει και το θέμα του backloading. Έχω όμως μια επιπλέον ερώτηση όσον αφορά αυτό το σημείο. Πώς θα συνδυάσουμε τις φιλοδοξίες αυτές με την απόλυτα θεμητή ανησυχία της βιομηχανίας. Και ιδιαίτερα τι εγγύσεις μπορείτε να δώσετε εσείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, σε αυτούς που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις, και το τονίζω αυτό, καλύτερες επιδόσεις στη βιομηχανία, προκειμένου να καταπολεμηθεί η λεγόμενη διαρροή διοξιδίου του άνθρακα και ιδιαίτερα μετά το 2020. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Παναλαμβάνω ότι έχουμε την πιο μεγάλη αγορά στον κόσμο. Και αναπτύσσουμε τέτοιες αγορές και αναπτύσσονται κι αλλού, Οι Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδειγματίζονται από αυτήν. Η Ελβετία. Στο μέλλον, μάλιστα, οι δικές μας αγορές θα πρέπει να συνδεθούν με τις υπόλοιπες στον κόσμο. Γι' αυτό και η ευθύνη που επομιζόμαστε είναι τεράστια για το πώς θα διαχειριστούμε αυτό το σύστημα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά να έχουμε η υπόψη μας και τα συμφέροντα της βιομηχανίας μας γιατί μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά που πρέπει να φροντίσουμε. Και για να τα φροντίσουμε πρέπει να έχουμε ένα βιομηχανικό τομέα με σημαντικό μέρος στην οικονομία μας που να είναι ανταγωνιστικός. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να συνεχίσουμε με το σύστημα αυτό δωρεάν ε, παραχώρησης δικαιωμάτων για να αποφύγουμε ακριβώς τη διαρροή διοξιδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο που είχαμε μέχρι τώρα από τις μελέτες της Επιτροπής διαπιστώσαμε ότι δεν μεταφέρθηκαν επιχειρήσεις αλλού, δεν μετεκαταστάθηκαν εξαιτία της αύξησης της τιμής άνθρακα. Μπορεί να αυξηθεί λίγο η τιμή. Τότε πρέπει να προστατεύσουμε τη βιομηχανία μας. Συνεπώς, στους πιο αποτελεσματικούς θα δώσουμε δωρεάν δικαιώματα. Πρέπει να σχεδιάσουμε ένα νέο σύστημα βέβαια, αλλά να λάβουμε υπόψη μας το πρόβλημα ορισμένων χωρών, οι οποίες εξαρτώνται πάρα πολύ από τον άνθρακα για τις δικές τους εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού και να δούμε τι εξαιρέσεις μπορούμε να προβλέψουμε για αυτές τις χώρες. Ώστε να στηρίξουμε τη... τον ηλεκτρισμό, τη βιομηχανία ηλεκτρισμού σε αυτές τις χώρες και παραγωγή ενέργεια γενικότερα. Έχουμε τεράστια ευθύνη, όντω όμω, να ανταμείψουμε αυτού που έχουν τι καλύτερε επιδόσει. Ευχαριστώ, κυρία Γκαρσία Πέρε. Ευχαριστώ. Κύριε Αρία Κανιέται, υποψήφιο επίτροπο για τι κλιματικέ αλλαγέ για την κλιματική δράση, ήσασταν υπουργό μια κυβέρνηση που ενέκρινε την νομοθεσία για τι ακτέ που ήταν όνειδο για ολόκληρη την Ευρώπη και θα ισοπεδώσει το, την, την φυσική μας κληρονομιά. Εσείς ως αρμόδιος υπουργός ήσασταν κατά των δεσμευτικών στόχων για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Τώρα βέβαια μας λέτε θα, ότι θα τους στηρίξετε τέτοιους δεσμευτικούς στόχους πέραν του χαρτοφυλακίου σας παραδεχτείτε ότι δεν μας κάνετε και τη ζωή εύκολη με κάποιες παράπλευρες πληροφορίες. Προσβάλλετε όλες τις γυναίκες. Επίσης, ε, για να συγκαλύψετε μια σαφέστατη σύγκρουση συμφερόντων, πουλάτε άρον-άρον τις μετοχές σας. Και μία μέρα πριν την ακρόαση, μόλις χθες, δηλώσατε ότι είχατε λάβει αμοιβέ από το Λαϊκό Κόμμα ενώ είχατε αποκρύψει εδώ και τρει μήνε την πληροφορία αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη δήλωση του πόθεν έσχε σα. Θεωρείστε ότι έχετε το ηθικό παράστημα για να γίνετε επίτροπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Ευρωβουλευτή. Έχω δύο σχόλια να κάνω. Εγώ ανέκαθεν και ως Υπουργό Περιβάλλοντος ψήφισε υπέρ των προτάσεων της Επιτρόπου Κόνι Χέλεγκαρτ και μπορείτε να δείτε τα πρακτικά του Συμβουλίου. Ήμουν ανέκαθεν στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπερψήφισα τις προτάσεις της. Ανήκα στην ομάδα για την πράσινη ανάπτυξη. Οι 13 ε, υπουργοί που ταχθήκαμε υπέρ των καθαρών ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και κατά των ορυκτών, ήμασταν εμείς. κατά των ορυκτών καυσίμων. Και τότε δεν ήμουν επίτροπο για καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πούλησα τις ε, μετοχές μου, όχι όπως είπατε, αλλά όταν έμαθα ότι με πρότειναν για Ευρωπαίο Επίτροπο. Με βάση τη διαφάνεια και τη συνέπεια. Και θέσπισα το νόμο για τις ακτές για να προασπίσω τα συμφέροντα πολλών Ευρωπαίων πολιτών που είχαν επενδύσει στην Ισπανία, είχαν αγοράσει κόπεδα στις Ισπανικές ακτές και μία ωραία πρωία τους λέει ένας νόμος ότι θα χάσουν την ιδιοκτησία τους. Όλα αυτά λοιπόν τα έκανα για να προστατεύσω τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό το έκανα. Και δεν έχω αποκρύψει τίποτα. Τίποτα δεν έχω αποκρύψει, κύριε Ευρωβουλευτή στο βιογραφικό μου αναφέρεται ότι διατέλεσα πρόεδρος της ε, Εκλογικής Επιτροπής. Είναι πολιτικό αξίωμα και μάλιστα δεν αμοιβόμουν γι' αυτό. Απλώς είχα έξοδα παράστασης. Και μάλιστα από την πρώτη στιγμή περιέλαβα αυτό το στοιχείο στη δήλωση πόθεν έσχες και στη δήλωση οικονομικών συμφερόντων προς την Επιτροπή. Από την πρώτη μέρα για να το γνωρίσει, να το αναλύσει και να το εγκρίνει η νομική υπηρεσία. Το δήλωσε και στην Ισπανική Εφορία. Πλήρωσα τους φόρους μου. Ήταν απόλυτα διαφανής όλες μου οι δραστηριότητες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφιο επίτροπε για τη δήλωσή σας. Ο κύριος Άσλι Φόξ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κύριε Κανιέτα. Εδώ είμαι. Θα μάθετε ότι δεν ενδιαφέρομαι για το τι κάνει ο κουνιάδος σας, ε, πώς βγάζει το ψωμί του. Υπάρχουν 248 σχέδια κοινού συμφέροντος ε, στα πλαίσια του τμήματος 10 της ε, δυνατότητας συνδέοντας την Ευρώπη. 5,8 δις ε, εκατομμύριο προπολογισμό τους για 5 χρόνια. 7 χρόνια, συγγνώμη. Τα περισσότερα λοιπόν δεν θα χρηματοδοτηθούν. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι κριτήρια θα χρησιμοποιήσετε για να αποφασίσετε ποια από αυτά τα προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν και ποια όχι. Ίσως ο πρόεδρος θα μπορούσε να παρακαλέσει τους σοσιαλιστές να σταματήσουν να συζητούν με τους συμβούλους τους. Επιπλέον, επιπλέον, πολλά λέγονται για προγράμματα για να βελτιωθούν η αγωγή φυσικού αερίου. Θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να βελτιωθεί και το ε, πλέγμα μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος στις χώρες μας. Θεωρώ ότι όλα τα προγράμματα της δυνατότητα, που δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθεί η Ευρώπη και να υπάρξουν διασυνδέσεις ως απόλυτη προτεραιότητα. Είναι αλήθεια ότι το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη έχει μόνο 5,8 δις. Ένα από αυτό που θα κάνω λοιπόν είναι όταν θα έχουμε την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου θα προτείνω ότι θα πρέπει αυτό να είναι προτεραιότητα της Ένωσης και στο πακέτο για τα 300 δις ε, που θα εφαρμόσουμε θα επιδιώξω να υπάρξει χρηματοδότηση για αυτά τα προγράμματα και επιπλέον όσο περισσότερα χρήματα μπορούμε να λάβουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στην επιλογή των προγραμμάτων ε, ενωσιακού συμφέροντος κάναμε κάτι που είναι σημαντικό. Δεν αποφασίζει η Επιτροπή τι πρόγραμμα θα προωθηθεί. Έχουμε περιφερειακές ομάδες με τις ρυθμιστικές αρχές, ε, τις επιχειρήσεις που λειτουργούν, διάφορα, το λειτουργούν το ενεργειακό πλαίσιο και διάφορους άλλους φορείς εμπλεκόμενους για να εκτιμήσουν ποια είναι τα καλύτερα. Και για μένα τα καλύτερα είναι αυτά που βοηθούν την διασύνδεση χωρών. Ούτως ώστε να αυξήσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης. Αυτά τα προγράμματα θα προωθήσουμε. Αλλά θα το αποφασίσουν οι περιφερειακές ομάδες. Πρέπει να ε, επαφιέμεθα στα περιφερειακά όργανα, όχι να αποφασίζει για αυτά τα, προγράμματα, τα προγράμματα ε, ενωσιακού συμφέροντο η Επιτροπή, αλλά είναι περιορισμένη η χρηματοδότηση. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και κατά την αναθεώρηση των προοπτικών θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερη χρηματοδότηση γιατί αυτά τα προγράμματα αξίζουν στήριξη. Ευχαριστώ πολύ. η, ο κύριος Χιράουτα Βιδάλ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή στήριξαν ε, πάρα πολύ την ε, διασύνδεση σε 10% στην Ευρώπη για τον ηλεκτρισμό και μάλιστα είπαν ότι για το 2030 θέλουν να είναι 15%. Η τήρηση του στόχου αυτού είναι το εμπόδιο για τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης. Και Μα δυσκολεύει επίση να πετύχουμε του στόχου μα ακόμα και για το 2020. Κάποιε χώρε μελή στις προσπάθειες που κάνουν για να πετύχουν του στόχου αυτού, ανέπτυξαν τις ε, ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας σε έναν βαθμό, χωρίς όμως να μπορέσουν να εξάγουν προς την υπόλοιπη Ευρώπη το πλεόνασμα ενέργειας που είχαν. Τι θα κάνετε λοιπόν για να συνδέσετε τους στόχους αυτούς με τους υπόλοιπους στόχους της κλιματικής ε, ατζέντα για να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο. Τι θα κάνετε με τις διασυνδέσεις αυτές και τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για να αυξήσετε την διασύνδεση ακριβώς αυτή. Απάντηση. Μία από τις προτεραιότητές μου θα είναι προσωπικά να δώσω όθηση σε όλα τα προγράμματα διασύνθεσης που είναι τόσο ανάγκη στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Βαλτική και τελειώνοντας με την Ιδρική Χερσόνησο και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα προγράμματα αυτά για το μέλλον. Αλλά για να έρθω στη συγκεκριμένη ερώτησή σας όσον αφορά την Ιβηρική, είναι αλήθεια ότι είμαστε ένας ενεργειακό θύλακας. Ότι έχουμε αναπτύξει ανανεώσιμες πηγές, αλλά με δύο προβλήματα. Τα δίκτυά μας δεν είναι αρκετά αφή ώστε να απορροφήσουν το πλεόνασμα που κατά καιρού υπάρχει και από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να εξάγουμε παρόλο που έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Πορτογαλία, ναι, στην Πορτογαλία ναι, αλλά στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να εξάγουμε. Ούτε στις γειτονικέ ε, χώρες, Ιταλία, Ενωμένο Βασίλειο, δεν ξέρω τι, ενώ αν είχαμε καλή διασύνδεση θα μπορούσαμε. Έχουμε κάνει κάποια βήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως προωθεί τον διάλογο ανάμεσα στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, ακριβώς ώστε τα προγράμματα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Και όπως λέει και η κυρία Δικαστήγιο, υπάρχει και ένα που έχει προχωρήσει κάπως περισσότερο. Μια διασύνδεση που περνάει από τα 400 στα 800 ΜΒ ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία. Τα άλλα καθυστερούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει πρώτα να πετύχει την πολιτική συμφωνία μεταξύ χωρών μελών ώστε να γίνει βιώσιμη η προσπάθεια αυτή και δεύτερον να βρεθεί η οικονομική στήριξη ώστε που είναι αναγκαία έτσι, για το ιδιωτικό τομέα ε, θέλει να έχει κάποιες εγγυήσεις για να προχωρήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως από την άλλη θέλει και αυτή τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Θέλουμε λοιπόν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο έτσι ώστε όλες οι άδειες να δίνονται σε μικρό χρονικό διάστημα. Θα αφοσιωθώ σε όλα αυτά και όχι μόνο για την Ιβυρική Χερσόνησο αλλά και για τις διασυνδέσεις ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κύριος Μύροσλαβ Ράνστορφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, στον ενεργειακό τομέα έχουμε κάποια φυσικά μονοπόλια αλλά το μέλλον της ενέργειας στην Ευρώπη ε, θα προβλέπει μια καλύτερη αξιοποίηση και ένα συνδυασμό των μεγάλων και των μικρότερων ενεργειακών δομών και υποδομών. Πώς θα εξισορροπήσουμε τις ε, μεγάλες με τις μικρότερες ενεργειακές δομές. Απάντηση. Πιστεύω ότι για να βρούμε την ισορροπία θα πρέπει καταρχήν να πατάξουμε τις μονοπολιακές πρακτικές. Αν υπάρχει κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, θα θέσω το ζήτημα στον αρμόδιο επίτροπο ανταγωνισμού για να διορθώσουμε τις περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Ο καλύτερος τρόπος λειτουργίας όμως είναι μία εσωτερική αγορά με τερματικούς σταθμούς. Δηλαδή, στο τρίτο ενεργειακό πακέτο θα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως όλα τα στοιχεία. Και φυσικά χρειαζόμαστε και νέα μέτρα για τα ευφύη δίκτυα, για τις διασυνδέσεις, για τις διασυνοριακές μεταφορές και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, γιατί θα πρέπει να δέσουμε τον καταναλωτή στο επίκεντρο του ενεργειακού συστήματος. Θέλουμε έξυπνους μετρητές, θέλουμε αποδοτικές οικιακές συσκευές με οικολογικό σχεδιασμό. Να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν τις καλύτερες ενεργειακές επιλογές. Θέλουμε ευφύ ενεργειακά δίκτυα, συμπερίληψη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και φυσικά πρόθεση της αυτοκατανάλωσης και αυτοπαραγωγής. Όλα αυτά θα τα επιτύχουμε και μια αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των διαφόρων στοιχείων με μια ολοκληρωμένη και διαφανή εσωτερική αγορά της ενέργειας. Είπα στην αρχή ότι βασικός μου στόχος είναι η συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς και θα ήθελα κατά το τέλος της θητείας να έχουμε μια εύρυθμη εσωτερική αγορά με διαφανή και οριζόντιο υπολογισμό των τιμών. Γιατί αν έχουμε μια ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά θα ενισχύσουμε και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε και μεγαλύτερη σύγκληση των τιμών προς τα κάτω. Αν συνεχίσουμε με κατακαιρματισμό τη αγορά και απομονωμένες αγορές, ούτε ανταγωνιστικότητα θα έχουμε, ούτε ε, υγιή ανταγωνισμό, ούτε χαμηλέ ενεργειακέ τιμέ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλώτ Τούρμες. Κύριε Κανιέτε, ως Ισπανός ε, Υπουργός Περιβάλλοντος, περιβάλλοντος, σας υπέρ της ε, ε υπέρ της ε, εισαγωγής ε, βρώμικων άμμων από τον Καναδά και επίσης θελήσατε τα παλιά πυρηνικά εργοστάσια να συνεχίσουν να λειτουργούν. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνούσατε ή ήσασταν υπερβολικά αδύναμος για να παρεμποδίσετε. Τώρα, ο Μιγγέλ Ντομέξολης δεν είναι κάποιος δεν είναι κάποιος ε, κουνιάδος σας. Είναι εδώ και 25 χρόνια μέλος της οικογένειάς σας αλλά και ε, ε, συνεταίρος σας επιχειρήσεις. Και επίσης εδώ και 13 χρόνια υπάρχει μια διαδικασία φόρο διαφυγής για μια επιχείρηση στην οποία παίζατε κύριο ρόλο. Πώς θέλετε με τέτοια δαμόκλειο σπάθη από πάνω σας να αναλάβετε τέτοια ευθύνη. κύριε Τούρμες. Δεν ξέρω πού τις έχετε αυτές τις πληροφορίες. Κοιτάξτε. Στην δήλωση συμφερόντων μου υπόθηκε ότι η... αναφέρεται ότι εγώ είμαι δικηγόρος. Έχω λοιπόν ε, διατελέσει σύμβουλο σε πολλές πανικές εταιρείες. Και ως υπουργό Περιβάλλοντος δεν έλαβα τις αποφάσεις αυτές. Στις κυβερνήσεις περνάει η άποψη κάποιου υπουργού κάποιε φορέ και άλλε όχι, όπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ μπορεί να κέρδισα όσον αφορά το backloading, αλλά έχασα άλλε μάχε. Αλλά τι μάχε πρέπει να τι δίνει κανεί. Ήμουν υπουργό περιβάλλοντο και επέβαλα μελέτε επιπτώσεων για όλα τα προγράμματα και μάλιστα τι πιο αυστηρέ που ποτέ υπήρξαν στην Ισπανία. Με, κριτήρι, με κριτέ, κριτήρια πάντα, πάντα παραλαμβάνω, επιστημονικά και τεχνικά, όχι πολιτικά. Και αναφέρεστε τώρα σε αυτά, αυτές τις άμμους πίσας. Και υπάρχει και το θέμα των βιοκαυσίμων εδώ. Και το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει κυρίαρχα τι θα γίνουν αυτά τα θέματα. Όταν θα υπάρξουν ε, κοινοτικές ρυθμίσεις που επιτρέπει να γίνεται κάτι, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να αντιπαρατεθεί. Η Ισπανία συμμορφούται με την Ισπανική νομοθεσία και αν δεν το κάνει θα υπάρξουν δράσεις και προσφυγές της ε, Επιτροπής ε, εναντίον της. Εγώ ως Επίτροπος θα σεβαστώ αυτήν την ε, νομοθεσία. Εάν γίνει πιο αυστηρή η κοινοτική νομοθεσία και απαγορευτεί η εισαγωγή άμμων πίσας, όπως συζητιέται αυτή τη στιγμή στον ΠΟΕ, τότε θα ε, το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή στην οδηγία για τα βιοκαύσιμα δεν γίνονται αυτές οι διακρίσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος David Coburn. Υποψήφια Επίτροπε, σαν ε, ένας ε, άντρας που γίνεται όλο και πιο διάσημος μιλώντας για τις πνευματικές ικανότητες των γυναικών, εγώ θα σας ρωτήσω για την ρήπανση και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλάει για την μείωση 40% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα όταν εκπέμπουμε 12% και το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο 2%. Δεν συμφωνείτε ότι με τον τρόπο αυτό θα ξοδευτούν φοβερά πολλά χρήματα για μέτρα μετριασμού της ε, ρήπανση που καταστρέφουν την οικονομία. Ενώ στην πραγματικότητα ό,τι και να κάνουμε τελικά για τις εκπομπές, οι εκπομπές θα αυξηθούν παγκοσμίω. Κάθε Κινέζος, κάθε Ινδός θέλει ένα ψυγείο, θέλει μια Φεράρι κτλ. Θα μπορούσα να σας ρωτήσω και για την οικογένειά σας. Πάντως διακόπτει το μικρόφωνο του ομιλητή ο πρόεδρος. Έληξε ο χρόνος σας, συνάδελφε, έληξε ο χρόνος σας. Παρακαλώ. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, να απαντήσετε παρακαλώ. Πρώτον, Νομίζετε ότι δεν χρειάζονται μέτρα. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Αυξάνει η θερμοκρασία του πλανήτη μας, πρέπει να περιοριστεί αύξηση αυτή στους δύο βαθμούς. Λέτε, γιατί να κάνουμε κάτι αφού εμείς ρηπαίνουμε κατά 11%. 40% μείωση των εκπομπών δεν έχει καμιά σχέση με το επίπεδο εκπομπών που έχουμε. Έχει να κάνει με την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε την ε, μείωση της αύξησης της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς. Και χρειάζεται κάποιο να έχει τον ηγετικό ρόλο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και αυτό που έχει αυτό τον ηγετικό ρόλο είμαστε εμεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κοπεχάγη και σε όλε τι διασκέψει κορυφή που έγιναν για αυτό το θέμα. Και πρέπει να συνεχίσουμε μέχρι το Παρίσι και να πείσουμε και άλλου να πάρουν τα ίδια μέτρα όπως παίρνουμε και εμείς. Γιατί δεν γίνεται να λέμε αφού δεν κάνουν οι άλλοι δεν κάνουμε ούτε και εμείς. Μα δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Η καταστροφή μας περιμένει αν δεν γίνει κάτι. Για να πείσουμε τους Κινέζους, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να προχωρήσουμε με φιλόδεξους στόχους για να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή, πρέπει να έχουμε ηγετικό ρόλο και να βρούμε και τα μέσα, γιατί αν θέλουμε μια πράσινη οικονομία, τότε θα γίνουμε ανταγωνιστικοί τότε θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Τέσσερα εκατομμύρια είναι σήμερα στην πράσινη οικονομία. Και είναι ο τομέας όπου έχουν χαθεί λιγότερες θέσεις απασχόλησης, που έχει ε, διατηρηθεί το επίπεδο και μέχρι το 2030 με τους φιλόδοξους στόχους μας θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης, εκατομμύρια. Αυτό είναι ο στόχο μα. Η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητά μα στην πράσινη οικονομία. Η χώρα σα είναι μια από τι πιο ανταγωνιστικέ στην πράσινη οικονομία, με νέα προϊόντα, νέες προδιαγραφές. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι ο στόχος που πρέπει να πετύχουμε. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό. Αν πιστεύουμε στο περιβάλλον, πρέπει να πιστέψουμε και σε αυτούς τους στόχους. Ευχαριστούμε κύριε Υποψήφια Επιτροπέ. Ο κύριος Μάρκος Πίπερ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Κανιέτα που με τόσο διαφανή και πλήρη τρόπο δηλώσατε τα οικονομικά σας συμφέροντα και νομίζω ότι και η δήλωση ότι λυπάστε για αυτά που είπατε για θέματα ισότητας γυναικών έπεισαν τους συναδέλφους. Θέλω να πω κάτι για την ενεργειακή απόδοση. Πολλά κράτη-μέλη έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα να επιτύχουν τους στόχους εξοικονόμησης που τους τίθενται γιατί είναι πολύ αναλυτικοί και γιατί είναι και ιδιαίτερα γραφειοκρατικοί. Κύριε Κανιέτε, πώς θα μπορούσαμε περισσότερη ευελιξία και με περισσότερα κίντρα να φροντίσουμε κάθε χώρα να αξιοποιήσει τα προτερήματά της, για παράδειγμα για τις ανανεώσιμες και για τα θέματα μείωσης του διοξειδίου του άνθρακος, ούτως ώστε κάθε χώρα να μπορεί να συμβάλλει επιτυχέστερα στην συνολική ε, εκπλήρωση των στόχων συνολικά της Ευρώπης. Ο κύριος Κανιάτα. Για να, για να επιτύχουμε τους γενικούς μας στόχους, πρέπει να γίνει σωστή κατανομή των στόχων ανά κράτος μέλος με ευφύ τρόπο λαμβάνοντα υπόψη τι δυνατότητες έχει κάθε κράτος μέλος και την κατάστασή του. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να γίνει και για το σύστημα εμπορίας, όπου υπάρχει ένα σύστημα καθορισμού προδιαγραφών, benchmarking, για το πώς δίδεται στόχο σε κάθε εταιρεία, εταιρεία και Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση κάθε χώρας και τις ανανεώσιμες. Δεν θα είναι δεσμευτική πλήρως η στόχη, αλλά θέλουμε δεσμεύσεις από διάφορα κράτη-μέλη, οπότε υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας με βάση τι ευκαιρίες, αλλά και τι ουσιαστικά δυνατότητες με βάση την μορφολογία του έχει το κάθε κράτος μέλος. Γιατί κάποιες δυνατότητες μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτύξουν ανανεώσιμες και άλλες όχι. Αλλά θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον 27% ανανεώσιμες. Και για την ενεργειακή απόδοση έχουμε πολλές δυνατότητες. Γιατί μπορούμε να εργαστούμε ακόμη και σε επίπεδο του κάθε πολίτη. Μπορούμε να ε, κάνουμε τις μεγαλύτερες οικονομίες στον τομέα των οικοδομών και στον τομέα της θέρμανσης. Να βοηθήσουμε λοιπόν ακόμη και τον κάθε πολίτη να επιλέξει τη μορφή θέρμανσής του για παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντικά μέσα με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, πολύ σημαντική ε, οδηγία, με την απόδοση των κτηρίων και επίσης θέλουμε να έχουμε και μετρητέ μετρητές όλα τα συστήματα. Εάν το επιτύχουμε θα έχουμε σε κάθε χώρα πολύ καλές εξοικονομίες ενέργειας, ε, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Μπορούμε να έχουμε 100 εκατομμύρια ευφυεί μετρητές στο μέλλον στην Ένωση και αυτό θα επιτρέψει σε κάθε καταναλωτή να είναι αποτελεσματικό. Ευχαριστώ κυρία Καβεσόν Ρουί. Ευχαριστώ. Κύριε Κανιέτε. Ε, τα λόγια έχουν μεγάλη δύναμη και σήμερα άκουσα πολλές υπερβολές που θα μπορούσα και να τις πιστέψω αν δεν είχα ήδη απείρα από την Ισπανία γιατί γνωρίζω τις πολιτικές σας και όντως σπεύσετε να διορθώσετε την δήλωση, ακόμη και το ήσασταν γερουσιαστής. Θα συλλητεύσετε την κυβέρνησή σας και θα ε, επιβάλλετε κυρώσεις ε, αν δεν, πληρώσει, δεν συμμορφωθούν τους στόχους του 2020. Εσείς καταστρέψετε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και με άδικο και ψευδό τρόπο μιλήσετε για ένα ε, έλλειμμα στο οποίο εσείς συμβάλλατε. Επίσης, ε, ε, θα δώσετε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για αυτοκατανάλωση και εκδημοκρατισμό της ενέργειας, ενώ για τα θέματα αυτά δημιουργήσατε πολλά εμπόδια στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Ξεκινώντας από το, από το πρώτο θέμα που είπατε, στην Γερουσία στην, και στην Ισπανική Βουλή δεν απέκρυψα κανένα στοιχείο. Όλα βγήκαν αυτά στον τύπο. Και τι έκανε η κυβέρνηση, τι ήταν το περίεργο που έκανε. Δημιούργησε ένα έλλειμμα στις, στην τιμολόγηση εξαιτία των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια υπερβολικό. Εσεί εσείς δεν το θεωρείτε ίσω υπερβολικό, αλλά τελικά την ύφη την πληρώνουν οι καταναλωτέ. Και μάλιστα αυτό εξαιτία μια ασφαλμένη πολιτική που οδήγησε σε έσοδα άνω του 20% που για σας μπορεί να είναι ε, σημαντικά, αλλά δεν είναι δεν... Ε, για σας μπορεί να είναι λογικά, αλλά δεν είναι λογικά για, το... για τα δημόσια οικονομικά. Ε, εμείς είμαστε υπέρ ε, μεγαλύτερης λειτουργίας της οικονομίας αγοράς και περιορισμού των κρατικών ενισχύσεων. Πάντως εγώ ως Επίτροπος θα εφαρμόσω την κοινοτική, την ενωσιακή νομοθεσία και θα επιβάλλω κυρώσεις και στην Ισπανική κυβέρνηση και σε οποιοδήποτε κράτος που θα παραβιάσει τους στόχους εφόσον είναι δεσμευτική. Αλλά μην ανησυχείτε, το 2013 η Ισπανία ήταν στο 16,1% και το 20% θα πάει στο 20%. Είναι από τις καλύτερες ε, ε, χώρες ε, με τις καλύτερες επιδόσεις στην ενέργεια. Δεν είναι ουραγός στην υλοποίηση των στόχων. Βέβαια, αν το 2020 δεν υλοποιηθούν οι στόχοι, θα πρέπει να εξετάσουμε τα αίτια της μη συμμόρφωσης. Επίσης, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να καλύψουν το χαμένο έδαφος ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι επιβάλλει κυρώσεις, αλλά να βοηθάει για την εφαρμογή τη ερωσιακής νομοθεσία. Βέβαια, αν κάποιε χώρε την παραβιάσουν, μην έχετε καμία εμφιβολία ότι θα υποστούν κυρώσεις. Εγώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα εκπροσωπώ την Ισπανία, αλλά το συμφέρον 500 εκατομμυρίων συμπολιτών μας. Αυτό είναι το καθήκον μου, αυτή είναι η δέσμευσή μου και αυτό θα κάνω αν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάνκαν είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κανιέτε, γνωρίζετε ότι η Σκοτία παράγει ενέργεια, είναι σημαντικός παραγωγός και υδρογοναθράκων και ανανάσιμων πηγών ενέργειας. Ελπίζω να έρθετε στη Σκοτία και να δείτε από μόνο σας πώς έχει η κατάσταση εκεί. Άκουσα τη στήριξή σας για το αβόριο δίκτυο, πολύ καλό αυτό. Θα θέλω όμως ένα χρονοδιάγραμμα και να μας πείτε και οικονομικά τι θα προβλεφθεί. Όσον αφορά την υδρορογμάτωση τώρα, δεν έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα ότι οι χώρες μέλη έχουν την αρμοδιότητα. Τι θα κάνετε όμως ώστε να εξακολουθήσουν να έχουν αρμοδιότητες οι χώρες μέλη για το ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά την ε, υδρογνωμάτωση μεταξύ άλλων, γιατί ξέροντας ότι και το φυσικό αέριο μπορεί να εμποδίσει την ε, μετακίνηση προς άλλες πηγές ενέργειας. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η Βόρεια Θάλασσα, η πρωτοβουλία για το δίκτυο αυτό, είναι κάτι βέβαια που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την διασύνδεση. Συνεπώς θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε να προσπαθήσω να δω πώς θα στηρίξουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και προγράμματα. Ξέρουμε ότι τα κονδύλια είναι περιορισμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει και με τη διασύνδεση στη Βαλτική. Θέλουμε και εκεί να βοηθήσουμε, γιατί όντω, όπω σα είπε η διασύνδεση πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η περιφερειακή προσέγγιση έχει τεράστια σημασία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά. Μπορούμε όμω να αρχίσουμε να τη φτιάχνουμε από το περιφερειακό επίπεδο, από περιφερειακές ολοκληρωμένες αγορές που θα αναπτύξουμε και θα τις συνδέσουμε μεταξύ τους ώστε να φτάσουμε σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά τελικά, που είναι και το τελικό αποτέλεσμα στο οποίο θέλουμε να καταλήξουμε. Υπάρχουν καλά παραδείγματα στις χώρες Μπενελούξ για παράδειγμα, που συμμετέχει και η Γερμανία. Υπάρχει αυτό το υπεράκτιο πλέγμα, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο την περιφερειακή προσέγγιση. Παντού, ώστε να διασυνδεθούν όχι μόνο είδη ενέργειας για να λύσουμε όσο γίνεται καλύτερα το πρόβλημα αυτό της ενέργειας. Όσον αφορά τώρα το σχεστολιθικό αέριο θα μελετήσω πώς λειτουργεί το σύστημα και θα υιοθετήσω νομοθεσία εφόσον προηγουμένως έχουμε δει τι θα γίνει στην Ευρώπη με την αρχική εμπειρία που θα έχουμε. Χωσέ Ιγνάτσιο Γαρία τώρα. Κύριε Κανιέτε. Στην γραπτή σας απάντηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλήσατε για την ανάγκη όλοι οι τομείς μεταφοράς να συμβάλλουν στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν πολλές ελλείψεις ε, και στις αερομεταφορές και στις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Θα πρέπει να ελέγξουμε τις, ε, τα καυσαέρια της ναυτιλίας και μετά να περάσουμε στον περιορισμό. Αλλά μην ξεχνούμε και τις αερομεταφορές η, ε, μόλις, η ρήπαση του περιβάλλοντος από τους δύο τομείς ε, μεταφορών έχουν σημαντικές ε, επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. Επίσης, οι διεθνείς αερομεταφορές έχουν εξαιρεθεί από το Διεθνές Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Σκοπεύετε να υιοθετήσετε πρωτοβουλίες πιο περιοριστικές και για τις θαλάσσιες μεταφορές και να μην δημιουργηθεί δυσμενής θέση της, ε, του ευρωπαϊκού κλάδου σε σχέση με τους υπόλοιπους. Επίσης τι θα γίνει με τους αερομεταφορές μετά το 2016, θα, δεν θα πρέπει να περιληφθούν και τα καυσαέρια και αυτού του τομέα για να συμβάλλει και αυτός μέχρι το 2016 στον περιορισμό των καυσαερίων. Σας ευχαριστώ. Πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί όλοι οι τομεί θα πρέπει να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και όντω, αυτή τη στιγμή έχουμε διαφοροποιημένη συμμετοχή των διαφόρων τομέων. Στην περίπτωση των μεταφορών και δι των αερομεταφορών, εμπίπτει στο σύστημα εμπορίας εκπομπών το ενδο, οι ενδοκινοτικές αερομεταφορές. Οι μεταφορές όμως ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα. Η ρύθμιση του προβλήματος αυτού θα πρέπει να λάβει υπόψη την ε, Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και το κατά πόσο θα μπορέσει αυτός ο οργανισμός να θεσπίσει μέτρα για την παγκόσμια αγορά. Αν το 2016 στην συνεδρίαση που θα γίνει στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας υποβληθούν θεσμευτικά μέτρα, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Αν όμως δεν καρποφορήσει αυτή η συνεδρίαση και δεν θεσπιστούν κάποια παγκόσμια μέτρα, αν η Παγκόσμια Οργάνωση Πολιτική Αεροπορία δεν τα καταφέρει να επιβάλλει δεσμευτικά μέτρα, τότε θα πρέπει να επανέλθουμε στην προηγούμενη οδηγία και θα πρέπει εμεί και εσεί να λάβω μία απόφαση για να δούμε αν θα την εφαρμόσουμε πλήρως, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, ή θα πρέπει να την τροποποιήσουμε. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε το 2016 για να δούμε τις εξελίξεις στην αρμόδια οργάνωση που ρυθμίζει τις αερομεταφορές. Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός θα εγκύψει και αυτό στο θέμα αυτό. Εμείς ε, έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα monitoring, ενημέρωσης και εξακρίβωση επαλήθευση για να δούμε ποιος ρηπαίνει. Ε, να δούμε αν κάποιος ρηπαίνει για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε κάποιους κανόνες, για να δούμε από πού προέρχονται οι εκπομπές στη, από την αυτιλία. Επίσης θα δούμε τι θα κάνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Αν δεν λάβει αποφάσεις, θα μπορούσαμε εμείς σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο να προτείνουμε κάποια μέτρα. Για τις δύο αυτές ε, μεταφορές, τις ναυτιλιακές και τις αερομεταφορές, περιμένουμε τους παγκόσμιους οργανισμούς να λάβουν κάποια μέτρα, γιατί είναι παγκόσμιο το θέμα και χρειάζεται μια παγκόσμια απάντηση. Κυρία Πιετικά είναι. Ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Με συγχωρείτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος αλλά κατάλαβα ότι δεσμεύεστε ιδιαιτέρως να καταπολεμήσετε την κλιματική αλλαγή που θεωρείτε ότι είναι πολύ σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα, ότι δεσμεύεστε να εργαστείτε για να υπάρξει αυτό το αποθεματικό για την ε, σταθερότητα της αγοράς για το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών και για άλλα μέτρα και θέλετε να υπάρχουν ευφιέστατα πανευρωπαϊκά δίκτυα, super smart και επίσης να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις και επίσης περισσότερες ανανεώσιμες. Θα ήθελα όμως λίγο περισσότερα σχόλια για αυτά. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιούμε ε, τις ε, ε, ενεργειακούς πόρους τρομερά πολλούς και θα χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερους. Με συγχωρείτε κυρία μου. Κύριε Πρόεδρε, δεν κατάλαβα. Αναφέρατε ένα ποσό. Τι ποσό, δεν κατάλαβα. Μία πρόταση. Παρακαλώ. Η ερώτηση. Πώς θα βοηθήσετε να έχουμε περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλές ε, δυνατότητες για να έχουμε περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, οι ανανεώσιμες. Μπορούμε να αναπτύξουμε τις ανανεώσιμες και επίσης να βοηθήσουμε μέσω νέα έρευνα και ανάπτυξη βιομηχανία να αξιοποιήσει περισσότερο τι ε, ανανεώσιμε. Έχουμε για παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά και την αιωλική ενέργεια. Υπάρχουν και άλλες μορφές ανανεώσιμες. Για παράδειγμα, υπάρχει η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Και, αυτή την, ε, και αυτόν τον κλάδο μπορούμε να αναπτύξουμε, άρα θα δημιουργώντας έτσι και ε, θέσεις εργασίας και μειώνοντας ε, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Επίσης περισσότερη ενεργειακή απόδοση. Να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας στις κατασκευές. Εργαστούμε μαζί με τον κλάδο για να το επιτύχουμε. Αυτή τη στιγμή ανανεώνουμε μόνο 1% των κτηρίων μας ε, των χρόνων. Αυτό είναι πολύ λίγο. Να περάσουμε στο 2. Αυτό δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, αυτό δημιουργεί πολλές πράσινες θέσεις εργασία. Επίσης, να χρησιμοποιήσουμε διάφορες συσκευές που θα μειώσουν την παραγωγή ενέργειας. Έχουμε τον οικολογικό σχεδιασμό των συσκευών. Θα μπορούσε να βοηθήσει και την ε, ε, η οικολογική σήμανση των συσκευών. Μπορούμε να αναπτύξουμε πολλούς τομείς. Καλύτερες τεχνικές καύσεις, ε, καλύτερες εγκαταστάσεις ε, στην, στα εργοστάσια για καλύτερη καύση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ περισσότερα. Πολλά μπορούμε να κάνουμε για να περάσουμε από την ενέργεια υψηλού άνθρακα στην ενέργεια χαμηλού. Η κυρία Σιμώνα Ποναφέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του κύριου Γιούγκερ, ακούσαμε για επιπλέον 300 δισεκατομμύρια επενδύσεις που θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς. Η Ευρώπη πρέπει όντως να επενδύσει και στον τομέα για τον οποίο εσείς είσαστε αρμόδιος. Οπότε θέλω να σας ζητήσω να μου πείτε αυτά τα 300 δισεκατομμύρια πού θα χρησιμοποιηθούν όσον αφορά τις ενεργειακές αλλαγές και τη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας λοιπόν σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να ενθαρρύνουμε και τη χρήση ανανόσιμων πηγών ενέργειας αλλά και την ενεργειακή επάρκεια. Και τι θα γίνει με τα δίκτυα, πώς θα τα αναπτύξετε περισσότερο απάντηση. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία με αυτήν τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποφεληθούμε δηλαδή από επενδύσεις στον τομέα ε, της ενέργειας και για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του κοινοτικού προϋπολογισμού, γιατί έχουμε ένα mainstreaming για όλα τα μέτρα, δηλαδή ώστε το 20% όλων των μέτρων να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση ανώσιμων πηγών αέρης κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να διασφαλίσει ότι οι χώρες μέλη θα χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνουν τα διαφορετικά ταμεία ώστε να κινητοποιήσουν πόρους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι πρώτες πληροφορίες λοιπόν που έχουμε από το πακέτο 2014-2020 είναι ότι τα πρώτα χρόνια 2014 καταρχήν, το ποσοστό χρήση των κονδυλίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι της τάξης του 12%. Τώρα όταν αρχίσουν και οι εταιρικέ συμφωνίες, το greening κτλ, πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε το 12%. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να βρει νέα συστήματα χρηματοδότησης προγραμμάτων, ομόλογα έργου και άλλες μορφές βοήθειας που θα κινητοποιήσουν ιδιωτικέ επενδύσει. Και στο πακέτο αυτό των 300 δισεκατομμυρίων, η ενέργεια, η ενεργειακή επάρκεια και ανανόσιμε πηγέ ενέργεια πρέπει να στηριχθούν ιδιαίτερα. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε και υπό την ε, Αντιπρόεδρο για την Ενεργειακή Ένωση αλλά και με τους υπόλοιπους επιτρόπους με εκείνον για την απασχόληση για παράδειγμα να κινητοποιήσουμε πόρους υπέρ της ε, ενέργειας. Με τον πρόεδρο Γιούγκερ, λοιπόν, με τα διευθυντικά ταμεία, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούμε να κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα υπέρ τη πράσινη οικονομία. Σε ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάβιο Τζανονάτ. Α, συγγνώμη. Πρώτα ο κύριος Πολ Ρούμπιχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω τον Επίτροπο εδώ στο Κοινοβούλιο μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε κάποιον που έχει εργαστεί στην πράξη γνωρίζει τα θέματα αυτά, μας φέρνει την εμπειρογνωμοσύνη. Είναι καλό να έχουμε τέτοιους που ήταν και στο Κοινοβούλιο τώρα σε επιτρόπους. Τι μέτρα θέλω να ρωτήσω μπορούμε να κάνουμε για την παραγωγή και για τους καταναλωτές. Πώς δηλαδή μπορούμε μέσω των καταναλωτών να έχουμε περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια ιδίω τα ιδιωτικά νοικοκυριά. Δηλαδή οι τιμές της ενέργειας να πέσουν γιατί ξέρετε ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα ενεργειακής και πώς θεωρείτε ότι η αποκέντρωση της παροχής ενέργειας μπορεί να βοηθήσει. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι στα πλαίσια των ευφυών τεχνολογιών θα ήταν δυνατόν να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πρέπει να αναπτύξουμε τα εφή δίκτυα και τους εφή. μετρητές. Είναι πολύ σημαντικό ο καταναλωτή να είναι στο κέντρο τη λήψη αποφάσεων. Πρέπει να μπορεί να επιλέξει πότε να καταναλώσει, πόσο να καταναλώσει, να γνωρίζει πάντα την ενημέρωση, αλλά με προστασία των δεδομένων. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Επίσης, αν αποφασίσει ο καταναλωτής να παραγάγει τη δική του ενέργεια μέσω αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις γι' αυτό. Πρέπει να υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο θα υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για να υπάρχουν κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο. Γιατί κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική προσέγγιση. Είναι ένα από τα θέματα για τα οποία έχει προστιθέμενη αξία η ευρωπαϊκή ρύθμιση. Πρέπει να ρυθμίσουμε πώς μπορεί να παραγάγει ενέργεια ο καταναλωτής, αλλά πώς θα συνδεθεί επίσης με το δίκτυο. Και μπορεί να χρειαστούν κάποιες επιδοτήσεις γι' αυτό και πώς θα ενταχθεί στο δίκτυο. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε. Πώς θα το κάνουμε. Και βεβαίως ε, υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που πάσχουν από ενεργειακή φτώχεια, που δεν έχουν πρόσβαση στην ενέργεια. Έχουμε και συστάσεις ε, του Φόρουμ Πολιτών γι' αυτό. Ποια πρέπει να τα μέτρα, ποιος είναι ο ορισμός των ενεργειακά ευαλώτων ατόμων. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από κράτος σε κράτος. Χρειάζεται κοινή προσέγγιση λοιπόν. Αλλά είναι σαφές ότι κάποια τμήματα του πληθυσμού έχουν μεγάλο πρόβλημα να πληρώσουν μια ενέργεια και θα πρέπει να βρεθεί καλύτερος τρόπος να τους βοηθήσουμε. Μέσω επιδομάτων ή μέσω ε, επιδοτήσεων για τα νοικοκυριά είναι περίπλοκα θέματα. Αλλά ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει οπωσδήποτε να τα δούμε και να προτείνουμε κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κανιέτε. Ο κύριος Φλάβιο Τζανονάτο. Ευχαριστώ. Εγώ έχω κάπως διαφορετική ερώτηση από αυτές που ακούσαμε επανειλημμένως. Πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότητα και ελαστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και χαμηλότερο κόστος. Αυτή ήταν η υπόσχεση που ακούσαμε, αλλά δυστυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Στην υδροελεκτρική ενέργεια, βασική πηγή του ενεργειακού μείγματος. Μία ενέργεια υδροελεκτρική ε, είναι παρούσα στην Ευρώπη πάνω από έναν αιώνα και αντιπροσωπεύει το 26% του συνόλου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και το 69% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην Ευρώπη, τα συστήματα παραχώρησης ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Κάποιες χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και άλλες προσπαθούν να επιβάλλουν μια απελευθέρωση του κλάδου. Δυστυχώς διακόπτει τον ομιλητή ο Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ένα από τα αποτελέσματα του τρίτου ενεργειακού πακέτου ήταν ότι έχουμε όλο και πιο ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές στα κράτη-μέλη. Επιπλέον, έχουμε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών. Βαίνουμε προς μία οδό ευρωπαϊκής ρυθμίσης μέσω των ενώσεων εθνικών αριθμιστικών αρχών και χάρη στην καλύτερη δικτύωση των φορέων των δικτύων και καλύτερο συντονισμό. Οδεύουμε προς μία εναρμόνιση. Βέβαια, όντως, ακόμη δεν έχουμε παρόμοιες καταστάσεις παντού και, και για την υδροελεκτρική ενέργεια έχουμε αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα. Πριν τη θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας, την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της αποτελεσματικής νομοθεσίας. Συμμερίζομαι την ανησυχία σας, αλλά θα πρέπει να αναλύσουμε αν θα επιφέρει προς τη θέμενη αξία μια πανευρωπαϊκή νομοθεσία ή απλώς θα επιτείνει τη γραφειοκρατία. Έχουμε αρμόδια αντιπρόεδρο που θα συντονίσει το το θέμα του εύνομοθετήν. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να θεσπίζουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία για να επιφέρουμε προστιθέμενη αξία και ε, πλεονεκτήματα που δεν μπορούν να επιφέρουν οι εθνικές νομοθεσίες. Ε, υπάρχουν βέβαια πολλά επιχειρήματα υπέρ της ολοκληρωμένης ε, εσωτερικής αγοράς, γιατί μια νέα αγορά, εσωτερική αγορά, θα έχει εναρμονισμένες τιμές, καλύτερη κυκλοφορία ενέργειας και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ανταγωνισμό ε, θεμητό. Φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε, όπως είπα, τις αρχές αναλογικότητας και επικουρικότητας. Είναι σημαντικές για να ε, έχουν εμπιστοσύνη οι πολίτες στο κύρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινωτικών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστούμε. Η κυρία Αγιούζο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε, Επίτροπε, όπως Μα είπε η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και είναι η αρμόδια για να το πει. Εδώ δεν πρόκειται για την προσπάθεια μόνο της αριστεράς η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει κόλλημα στη διαδικασία και επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια. Εσείς είσαστε αρμόδιος για να αναλάβετε το χαρτοφυλάκιο που σας έχει προταθεί. Εδώ θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό είσαστε ακριβώ ο κατάλληλο άνθρωπο. Λοιπόν, σε σχέση με τι προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, φυσικό αέριο και τα προβλήματα που υπάρχουν σε διάφορε ευρωπαϊκές χώρες, εσείς πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή πολιτική, η εξωτερική ενεργειακή πολιτική τη Ευρώπη τα επόμενα χρόνια και τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει στα εξωτερικά σύνορα και τι νέε διόδου μπορούμε να βρούμε, τι νέε διαδρομέ μπορούμε να βρούμε για την ενεργειακή μα κάλυψη. Απάντηση. Επιθυμία μου θα ήταν το South Stream, η διαδρομή αυτή, να αρχίσει να λειτουργεί. Γιατί έτσι έχουμε μια απόλυτη εγγύηση ότι τηρείται η κοινοτική νομοθεσία. Αυτό είναι το επιθυμητό. Αλλά τον ε, νότιο διάδρομο πρέπει να τον ε, προωθήσουμε και να φροντίσουμε ο ιδιωτικός τομέας να τον ενισχύσει. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε για τη διασύνδεση των βαλτικών χωρών, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, και να υπάρξει συγχρονισμός του ενεργειακού συστήματος της Βαλτικής με το ευρωπαϊκό, κάτι το οποίο κοστίζει, αλλά είναι αναγκαίο γιατί διασφαλίζει ενεργειακή ανεξαρτησία. Πρέπει επίσης να βασιστούμε στις ε, ντόπιε πηγές ενέργειας, όσο γίνεται περισσότερο. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό, να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση, γιατί τότε θα αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε λιγότερο, θα εξαρτώμεθα λιγότερο από αυτούς που μας ε, εξάγουν φυσικό αέριο. Το ευρωπημένο αέριο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε να δημιουργηθούν hubs στη Νότια Ευρώπη. Πολλές δυνατότητες υπάρχουν συγχρόνως, αλλά να μην εξαρτώμεθα από μια ενιαία πηγή, από μια ενιαία πρόσβαση. Για τελειώς θα δυσκολευτούμε από το φθινόπωρο. Όλοι μπορούμε να αγοράζουμε περισσότερο και πρέπει να ενωθούμε σε αυτό. Η Ευρώπη έχει μεγάλη αγοριστική δύναμη σε αυτό το τομέα στην ενέργεια και εγώ ως Επίτροπος, εάν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φτιάξουν πλατφόρμες κοινέ για την αγορά ενέργειας και τηρούν τις ρυθμίσεις του ΠΟΕ και τους κανόνες ανταγωνισμού, τότε θα το στηρίξω. Η Ευρώπη μπορεί να βελτιώσει πάρα πολύ τη θέση της σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε υποψήφι Επίτροπε. Η κυρία Γιούτε Ρούτελαντ. Κύριε Κανιέτε, το χαρτοφυλάκι όσος ε, λέγεται ότι πρέπει να είστε επικεφαλής των, προσπαθειών, των προσπαθειών για το κλίμα και τις ενέργειες για τις διαπραγματεύσεις. Μας αναφέρατε τους στόχους για τις εκπομπές, αλλά θέλουμε να μας μιλήσετε και για την ενεργειακή ασφάλεια. Θα προσπαθήσετε να υπάρχουν δεσμευτικοί φιλόδοξοι στόχοι για τα κράτη-μέλη, για πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας και για ανανεώσιμες. Συζητήσαμε επίσης και θέματα ναυτιλίας. Θα αγωνιστείτε ουσιοδός να σημειωθεί πρόοδο στο θέμα αυτό για γιατί η απάντησή σας ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που θα χαράξουν νέους δρόμους στον τομέα αυτό. Πολλές γυναίκες και κοπέλες θέλουν να μας πείτε επίσης τι πιστεύετε για τις διανοητικές διανοητικές τους Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε. Για τα θέματα ναυτιλίας. Το θέμα με την ναυτιλιακή πολιτική είναι ότι πρέπει να ξέρουμε τι εκπομπές έχουμε πριν ε, προτείνουμε ανώτατα όρια ελέγχου μειώσεων. Πρέπει να ξέρουμε τι επίπεδο εκπομπών έχουμε. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει ένα ευφυές σύστημα παρακολούθησης υποβολής εκθέσεων για να δούμε ποιες είναι αυτές οι εκθέσεις και για να ελέγξουμε πόσες είναι. Μόλις έχουμε τα στοιχεία αυτά θα είμαστε σε θέση να λάβουμε αποφάσεις. Αλλά επειδή το πρόβλημα των ε, θαλασσίων μεταφορών είναι πλανητικό, διότι όπως ξέρετε τα μεγάλα πλοία ε, διασχίζουν τον κόσμο, πρέπει να υπάρχουν συνολικά μέτρα για τα πλοία από ε, κάποιες διαστάσεις και πάνω. Οπότε ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας, IMO, στην επόμενη συνάντησή του θα δει αν θα ληφθούν αποφάσεις για το θέμα αυτό ή όχι. Εάν δεν τις λάβει, θα τις λάβουμε εμείς. Διότι μας ενδιαφέρει τα πλοία μας να είναι αποτελεσματικά ενεργειακά και να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους. Δεύτερον, για τους στόχους ενεργειακής ε, ασφάλειας. Για την ασφάλεια, ασφάλεια της προμήθειας. Πρέπει να εργαστούμε σε όλα τα μέτωπα, ούτως ώστε όλες οι χώρες να έχουν εγγυημένη αυτή την ασφάλεια προμήθειας. Έχουμε το πρόβλημα με την Ουκρανία, γεωπολιτική σύραξη. Αλλά η αστάθεια μπορεί να υπάρξει, για παράδειγμα, στην Νότια Μεσόγειο, μπορεί επίσης ε, σε άλλες συγκυρίες να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα πρέπει οι ροές να είναι αντιστρέψιμες, να έχουμε συστήματα, συστήματα διασύνδεσης με αντιστρέψιμες ροές και συστήματα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και αλληλεγγύης ανά Η ασφάλεια προμήθειας είναι πολύ σημαντική για μια Ευρώπη ανταγωνιστική στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χένα Βιρκούνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Κανιέτε. Όπως ξέρουμε, η συζήτηση αυτή τη στιγμή και η διαδικασία λήψη αποφάσεων για, για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές ε, έχει ε, χαράξει ένα σύνορο μεταξύ τους ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί επειδή δεν έχει μια γενική επισκόπηση κατάσταση. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την ενέργεια από το περιβάλλον. Θα πρέπει να φροντίσουμε για την ανταγωνιστικότητά μας και να εξασφαλίσουμε πρόσβαση ε, των επιχειρήσεων σε, προσιτή, σε ενέργεια σε προσιτές τιμές αλλά και φιλοπεριβαλλοντική. Ο πρόεδρος Γιούγκερ συνένωσε αυτά τα δύο θέματα στο δικό σας χαρτοφυλάκιο για να διορθώσουμε το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει ε, το έργο της το Νοέμβριο. Κύριε Κανιέτε, ήδη μας είπατε πόσο σημαντική είναι η πράσινη φιλοπεριβαλλοντική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ρωτώ λοιπόν ποια κατά τη γνώμη σας θα είναι τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Δυστυχώς διακόπτει ο πρόεδρος στα μέσα της ερώτησης. Αν καταλάβατε κάτι απαντήστε, λέει ο πρόεδρος. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την εξασφάλιση της φιλοπεριβαλλοντικής ανάπτυξης, της πράσινης ανάπτυξης. Το πιο σημαντικό που θα πρέπει να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βεβαιότητα και ασφάλεια δικαίου. Μόνο με ασφάλεια δικαίου θα προσελκύσουμε επενδυτέ για να επενδύσουν σε προγράμματα και σχέδια και σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Θα πρέπει να ξέρουν οι επενδυτέ ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο και με το που θα συμφωνηθεί στο, τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο το πακέτο για το 2030 θα πρέπει να ξεκινήσουμε σε συνεργασία με το περιβάλλον, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγγνώμη, συζήτηση για όλους τους κανόνες για να δούμε πώς θα αναπτύξουμε και θα μεταρρυθμίσουμε ε, την, το σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών, την ε, οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, τις δεσμεύσει των κρατών μελών για τις ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας, το νέο σύστημα διακυβέρνησης και ούτω καθεξής, ώστε πολύ σύντομα να γνωρίζουν όλοι οι βασικοί μα εταίροι στον κόσμο ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Επίσης, οι, πολι... οι κλιματικές αλλαγές θα πρέπει οριζόνται να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τι πολιτικές των διαρθρωτικών ταμείων. Και με τα κονδύλια που έχουμε προσημειώσει στο πακέτο Juncker θα μπούμε στο σωστό δρόμο για την πράσινη ανάπτυξη. Γιατί θα έχουμε επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς τομείς. Ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και στις διασυνδέσεις. Θα υποβληθούν πολλά σχέδια και προγράμματα για τις διασυνδέσεις. Έτσι θα εντατικοποιηθούν οι δραστηριότητε και θα γίνει πραγματικότητα η πράσινη ανάπτυξη. Τεράστιες ευκαιρίες και δυναμικό. Να γίνουμε πρωταγωνιστές σε βιομηχανίες με χαμηλή χρήση άνθρακα, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει εμείς να δώσουμε το παράδειγμα και ο υπόλοιπος κόσμος θα μας ακολουθήσει. Δεν θα πρέπει να ε, ζητούμε μόνο οι υψηλότερε δεσμεύσεις στο Παρίσι, αλλά να αναπτύξουμε και νέες τεχνολογίες. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη που σας κόβω, αλλά είναι οι δημοκρατικοί κανόνες. Αυτοί να τηρούμε το χρόνο. Η κυρία Τερέσα Γκρίφιν είναι η επόμενη. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Πουλήσατε βέβαια τι μετοχέ σα πρόσφατα. παρόλα αυτά, ήσασταν πρόεδρο των εταιριών αυτών και δημιουργήσατε στενέ διασυνδέσει με την πετρελαϊκή βιομηχανία. Πώ θα είσαστε αντικειμενικό λοιπόν στο μέλλον, στο ρόλο σας απέναντι στη βιομηχανία. Δεύτερον, σε πολλά μέρη της Ευρώπης η ενέργεια κοστίζει όλο και παραπάνω κάτι που πιέζει πάρα πολύ τους πιο ευάλωτους και τους πιο φτωχούς της κοινωνίας μας. Κανένας πολίτης δεν πρέπει να είναι αναγκασμένος να διαλέξει κατά πόσο θα ζεσταθεί ή θα φάει. Τι συγκεκριμένες προτάσεις λοιπόν θα υποβάλλετε ως Επίτροπος για να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό της ενεργειακής ένδυας. Τέλος, μπορείτε να διευκρινίσετε λιγάκι τα σχόλιά σας στο όταν λέτε ότι είναι δύσκολο να συζητήσουν άντρες με γυναίκες επειδή έτσι η πνευματική υπεροχή των ανδρών είναι σε βάρος των γυναικών. Απάντηση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συζητάω με γυναίκες. Είπα εξάλλου στην αρχή ότι ήταν λάθος το σχόλιο μου αυτό και ζήτησα συγγνώμη. Ήτανε σφάλμα. Ζήτησα συγγνώμη, αλλά βλέπετε ότι συζητάμε, το συζητάμε χωρίς πρόβλημα. Τώρα για τις πιο σχετικές ερωτήσεις σας. Ανεξάρτητος ήμουνα πάντα στη ζωή μου. Και όντω ήμουν ιδιοκτήτης αυτών των πιο διάσημων μετοχών της Ευρώπης, έτσι. Αλλά ήμουνα και στο Green Group εκείνη την εποχή ήμουνα υπέρ της πράσινης ενέργειας. Αυτή ήταν η θέση μου. Και ζητούσα φιλόδοξους κλιματικούς στόχους και στήριζα την καθαρή ενέργεια. Το έκανα στο παρελθόν, θα το κάνω και στο μέλλον. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα συμφέροντά μου και αν υπάρξει κάποια στιγμή τέτοιο θέμα υπάρχει ο κώδικας διοντολογίας των επιτρόπων. Βάσει αυτού θα πορευθώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για τους πιο ευάλωτους συμπολίτε μας. Πολύ σημαντικό. Έγιναν προσπάθειες για ένα κοινό ορισμό, για μια κοινή προσέγγιση. Το θέμα λοιπόν σήμερα είναι μέσα στην ενεργειακή μας πολιτική θα ασχοληθούμε με αυτό ή σε διάφορες πολιτικές, κοινωνικές κλπ. Στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής η καλύτερη προσέγγιση είναι να έχουμε ευφύς μετρητές ώστε να μπορούμε να πετύχουμε και καλύτερη τιμολόγηση, να κοστίζει λιγότερο η θέρμανση και να δίνουμε προτεραιότητα όταν ένα κράτος μέλος στηρίζει νέα κτίρια κτλ. να μπορεί να στηρίξει και το πιο ευάλωτο πληθυσμό ώστε να κοστίζει λιγότερο η ενέργεια, φροντίζοντα δηλαδή για καλύτερη μόνωση των κτηρίων κτλ. Έχουμε πάντως πολλές δυσκολίες και χρειάζεται ακόμα στήριση πρέπει να το σκεφτούμε ακόμα περισσότερο πώς θα δίνουμε αυτή τη στήριξη. Είναι ζωτική σημασία στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Φρανσουάς Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Απλή γυναίκα είμαι και θεωρώ παρόλα αυτά ότι ο κύριος Γιούνκερ είχε δίκιο να σας αναθέσει αυτό το χαρτοφυλάκιο γιατί ε, είστε απόλυτα εξοικειωμένο ε, με τα θέματα του χαρτοφυλακίου σα Και χαίρομαι για τον αποφασιστικό και κατηγορηματικό σα τόνο που δείχνει επιθυμία να πείσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στι προηγούμενε ακροάσεις δεν είχαμε πάντα την αίσθηση ότι ο συνομιλητή μα είναι απόλυτα ικανό και επαρκή για τη θέση όπω εσεί. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, σε μια οικονομία χωρί άνθρακα, ε, η διαδικασία δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Βέβαια, στις 8 Ιουλίου του 2014, η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αφιερώσει 300 εκατομμύρια ευρώ μόνο σε ένα θέμα, το θέμα της, δέσμευση δέσμευσης και αποθήκευση άθρακα. Θα το αναπτύξετε αυτό το πρόγραμμα και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ουδέποτε δεν μιλήσατε για την αποθήκευση ενέργειας. Αυτό είναι, αυτό και είναι σημαντικό θέμα. Έχετε το λόγο κύριε Κανιέτε. Θεωρώ ότι το θέμα της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο άνθρακας ε, για πολύ καιρό θα μείνει παρόν στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα και μεσοπρόθεσμα ε, ο άνθρακας ε, και ο λιγνίτης έχουν σημαντική μαρουσία στο ενεργειακό μείγμα πολλών χωρών και για να επιτρέψουμε στις χώρες αυτές να χρησιμοποιήσουν αυτόχθονες εχώριες πηγές ενέργειας, άνθρακα και λιγνίτη δηλαδή, θα πρέπει να αναπτύξουμε προγράμματα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Βέβαια δεν φτάσαμε ακόμη στη φάση εμπορίας διάθεσης στην αγορά. Αλλά από τα έξι προγράμματα που ενέκρινε η Διεύθυνση Ενέργειας από τα έξι προγράμματα που επέλεξε τέσσερα ε, έχουν ε, ε, αποτύχει, αλλά δύο έχουν μεγάλες πιθανότητες να φτάσουν στην αγορά. Έχουμε και το πρόγραμμα NERSIN 1 με 300 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση για την ανάπτυξή του. Και πολλά κρατημέλη είναι υπέρ αυτού του σχεδίου. Κυρίως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει αυτό το Nursing 1. Υποστηρίζει τέτοια προγράμματα και θα προσφέρουν και τεχνολογία που θα την αξιοποιήσουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εγώ θα υποστηρίξω τέτοια προγράμματα, την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων και την εξασφάλιση χρηματοδότησης τους. Γιατί σίγουρα ο άνθρακας είναι σημαντική πηγή ενέργειας. Τώρα, για την αποθήκευση ενέργειας. Οι συσσωρευτές είναι δαπανηροί, δεν είναι και πολύ αποτελεσματικοί, δεν είναι εύκολη η αποθήκευση ενέργεια. Έχουμε βέβαια κάποια προγράμματα που προτάθηκαν για αποθήκευση μέσω συστοιχειών. Θα το δούμε. Ίσως είναι χρήσιμα και για τη θέρμανση. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό. Αλλά χρειάζεται έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη γιατί ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε επίπεδο ώστε να μπορούμε να αξιοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες. Ο Γιολάινεν. Μια πολιτική, μια προσωπική ερώτηση. Επανειλημμένα είπατε ότι ως Επίτροπος θα είστε ουδέτερος σε σχέση με τις πηγές ενέργειας για την υδρογμάτωση, την εξόριξη πετρελαίου, τον άνθρακα. Σωστό είναι αν είστε Επίτροπος Ενέργειας, αλλά η Επίτροπος Περιβάλλοντος δεν είναι λάθος. Εάν θέλουμε να είμαστε παράδειγμα, πρέπει να φύγουμε από τις παλιές ενέργειες, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να τις περιορίσουμε. Οπότε έχετε μια πολιτική σύγκρουση συμφερόντων. Και ε, θεωρώ ότι συχνά μπορεί να είστε στη λάθος πλευρά όταν τα λόμπι είναι πολύ ισχυρά. Προσωπική ερώτηση. Προσωπική ερώτηση μετά την πολιτική. Προσωπική. Ε, αναφερθήκατε στον κώδικα δεοντολογίας όπου λέει ότι και προσωπικά και οικογενειακά πρέπει να είστε χωρίς συμφέροντα. Ισχύει ότι ο γαμπρός σας είναι ενεργός στην βιομηχανία πετρελαίου. Και τι θα πείτε στον ε, κύριο Γιούνκερ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, παρακαλώ. Κύριε Λάινεν, όταν ε, μιλούσα για την ε, πυρηνική ενέργεια και την υδρορογμάτωση, είπα για την πυρηνική ενέργεια η υποχρέωσή μου είναι να υπάρχει πυρηνική ασφάλεια, να διασφαλιστεί πυρηνική ασφάλεια με βάση τι υψηλότερε προδιαγραφέ ασφαλεία για του Ευρωπαίου πολίτε. Αυτή είναι η δέσμευσή μου. Για την υδρορογμάτωση είναι αποφάση των κρατών μελών. Η Επιτροπή έκανε συστάσει. Αν χρειαστεί, θα προχωρήσουμε και στην ε, επιβολή κανόνων. Αν χρειαστεί. Τώρα για τη σύγκρουση συμφερόντων. Κοιτάξτε, θα είμαι απόλυτα διαφανή. Θα δείτε και στην ιστοσελίδα μου, εάν γίνω επίτροπο, όλε τι συναντήσει που έχω κάνει με όλα τα άτομα, τι εταιρείε, τα λόμπι, Όλα, όλα θα τα βλέπετε, θα δείτε με ποιον συναντώμε και γιατί. Θα είμαι απόλυτα διαφανής. Και σας είπα ότι έχω ήδη πει. Πούλησα τις μετοχές μου παρά το ότι δεν συνιστούσαν σύγκρουση περιβάλλοντος γιατί σας είπα τι εταιρεία ήταν. Ήταν μια εταιρεία επιμελητίας και αποθήκευσης. Ούτε η ε, γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου, ούτε εγώ έχουμε την παραμικρή μετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία. Και εγώ θα εργαστώ για τα συμφέροντα των Ευρωπαίων. Θα αναπτύξω καθαρέ ενέργειε και για την ε, περίπτωση του άνθρακα. Ανησυχώ, γιατί υπάρχουν χώρε όπω η Πολωνία που έχουν ουσιώδε πρόβλημα. Πρέπει να αναπτυχθεί η δέσμευση και αποθήκευση για να μπορέσουν να διατηρήσουν την παραγωγή ενέργειας μέσω του άνθρακα. Θα στηρίξω λοιπόν τις πιο αποδοτικές τεχνολογίες γιατί το ενεργειακό μείγμα δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Ο άνθρακας θα συνεχίσει να είναι πολύ σημαντικός. Στο μέλλον να περάσουμε σε καθαρότερες ανανεώσιμες. Αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να γίνει αυτό και εντωμεταξύ θα υπάρξει νομοθεσία για να έχουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές για την πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Και Τελευταίος, ο Herbert Royal. Παρά την ε, εντύπωση που προσπαθούν να δημιουργήσουν ορισμένοι, δεν είναι εκπρόσωπος των πετρελαϊκών εταιριών, αλλά ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας που είχε μια εταιρεία με 50 εργαζόμενους, 50, 5-0. Καμία σύγκρουση συμφερόταν, αλλά παρόλα αυτά σωστά πούλησε και εκείνος και τα παιδιά τους τις ε, μετοχές τους. Δεν ήταν αναγκαίο να το κάνουν. Τώρα μιλάτε για τη γιαγιά του, τον κουνιάδο του. Δεν νομίζω ότι το παρακάνετε. Όλα αυτά δεν νομίζω ότι είναι δίκαια. Δεύτερον, δεύτερον, δεύτερον. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις παρακαλώ. Κύριε υποψήφια επίτροπε. Πώς, πώς, είπατε ότι μπορείτε πολλά να κάνετε, αλλά Πώς θα συνδυάσετε την ασφάλεια και τον ανταγωνισμό και την ε, πολιτική για το κλίμα. Τι μπορεί να κάνει ο Επίτροπος για να μην έχουμε διακοπή της παροχής φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπο. Ευχαριστώ κύριε Ρόιλ για το τελευταίο τμήμα της ερώτησής σας. καλοκαίρι έγιναν διάφορες δοκιμές αντοχής μετά την κρίση με την Ουκρανία για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα με υπόθεση εργασίας ότι θα σταματούσε η ροή φυσικού αερίου. Και ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι δοκιμές για να δείξουν ότι αυτές οι αμφίροπες ροές υπάρχουν, οι αμφίδρομες, ότι έτσι θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα. Στο μέλλον όμως, Πρέπει να διαφοροποιήσουμε οπωσδήποτε τις πηγές ανεφοδιασμού μας. Με το νότιο διάδρομο, με ανάπτυξη καλύτερων διευκολύσεων hubs, λιμένων, αλλά προκειμένου να είναι ανταγωνιστική βιομηχανία αυτή, πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω, δίνοντας δωρεάν δικαιώματα, αλλά και με μια εσωτερική αγορά που να λειτουργεί καλά μια εσωτερική αγορά, δηλαδή όπου να υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός και όπου οι τιμές είναι ίδιες ουσιαστικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου θα έχουμε διαφοροποίησει τις πηγές ενέργειας και θα χρησιμοποιούμε περισσότερο τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη χρήση της ενέργειας για να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να αναπτύξει νέες τεχνολογίες και όσον αφορά την δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Θα αναπτύξουμε επίσης καλύτερες τεχνολογίες για τις αναλλακτικές πηγές ενέργειας και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Η ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή συνδέονται και θα αποτελέσουν μια σημαντική ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ υποψήφια Επίτροπε, για τις απαντήσεις σας. Έληξε λοιπόν το τμήμα ερωταπαντήσεων της ακροασής μας. Ε, παρακαλώ μια σύντομη παρέμβασή σας κύριε υποψήφιε Επίτροπε για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ευρωβουλευτές, κυρίες και κυρίους. Σας ευχαριστώ πραγματικά όλους για τις ερωτήσεις σας. Χωρίς καμία εξαίρεση. Προσπάθησα να απαντήσω όσο μπορούσα καλύτερα. Αυτό που μπορώ να σας εγγυθώ είναι ότι έχω τον ενθουσιασμό και έχω και τη θέληση να αναπτύξω περισσότερο τις αρμοδιότητες που μου ανέθεσε ο κύριος Γιούνκερ εφόσον επιβεβαιωθώ στο χαρτοφυλακιό μου. Ειλικρινά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη. Πιστεύω ότι θα είμαστε στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και θα πετύχουμε εμπορικές συμφωνίες οι οποίες δεν θα μας οδηγήσουν σε μετεκατάσταση των βιομηχανιών μας εκτός Ευρώπης. Και πιστεύω πραγματικά ότι εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε ικανοί να έχουμε ενεργειακά δίκτυα απόλυτα διασυνδεδεμένα και μια εσωτερική αγορά που να λειτουργεί καλά. Γι' αυτό βασίζομαι στο συντονισμό με την Αντιπρόεδρο αλλά και με τους Αντιπροέδρους για την απασχόληση και στη συνεργασία με τους υπόλοιπους επιτρόπους. Πάνω απ' όλα όμως, κυρίες και κύριοι, θέλω να μπορώ να βασιστώ στην συνεργασία μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι απαραίτητο και το ξέρω αυτό από την εμπειρία μου ως Ευρωβουλευτής. 13 χρόνια ήμουνα στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω Ποιε είναι οι επιθυμίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν λοιπόν έχω την εμπιστοσύνη σα να ξέρετε ότι θα είμαι επιμονή μου βάσεω στη διάθεσή σα. Θέλω να υπάρχει διαφάνεια απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω και δεσμεύομαι να προχωρήσω σε μελέτες αντικτύπου για κάθε πρότασή μου. Πολύ σοβαρές μελέτες και πολύ αυστηρές και για τις οικονομικές επιπτώσεις και για τις κοινωνικές επιπτώσεις και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θέλω επίσης η διαβούλευση με τους πολίτες να είναι σε μόνιμη βάση και να είναι σοβαρή η διαβούλευση αυτή. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργάζεται μαζί μου από την αρχή της κάθε πρωτοβουλίας. Έτσι, χέρι-χέρι θα προχωρήσουμε στις σημαντικές δεσμεύσεις που πρέπει να αναλάβουμε, διότι οι στόχοι μας είναι περίπλοκοι. Πρέπει να έχουμε ηγετική θέση στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να μιλάμε με μία μόνο φωνή. Πρέπει να διαπραγματευόμαστε με μία φωνή όταν μιλάμε για την αγορά εκπομπών. Πρέπει να δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι παραπάνω από 28 χώρες μαζί. Και έχω τη στήριξη δύο γενικών διευθύνσεων που τις γνωρίζετε πολύ καλά. Η Επιτροπή Ήτρε συνεργάζεται με τη μία και η Επιτροπή Ένβη με την άλλη. Υπάρχουν εξαίρετοι αξιωματούχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν τις καλύτερες δυνατότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα καλύτερα προσόντα. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε συντονισμένα. Ξέρω ότι ορισμένοι από εσά έχουν επιφυλάξεις όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο αυτό. Αλλά πιστεύω ότι αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για όλους, με επιλογές καλά ισορροπημένες, φιλόδοξες πάντα. Και εννοείται, είμαι σίγουρος ότι αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά, θα δώσουμε και απάντηση στα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επόμενες γενιές το αξίζουν. Αξίζουν ένα περιβάλλον καλό, βιοπικιλότητα, δεν πρέπει να θέσουμε τις επόμενες γενιές σε κίνδυνο όσον αφορά τα θέματα αυτά. Τα 5 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη επίσης απαιτούν μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θέλουν οικονομική ανάπτυξη. Θέλουν οι περιβαλλοντικές μας προδιαγραφές να συνοδεύονται από την ανάπτυξη αυτή. Είναι μια ισορροπία δύσκολο να επιτευχθεί. Δεν είναι εύκολη. Και το ξέρω. Γι' αυτό και δεσμεύομαι απέναντί σας να προχωρήσω προς τους στόχους αυτούς με τη δικιά σας συνεργασία, με τη συνεργασία όλων. Είμαι συνεπώς στη διάθεσή σας εφόσον ε, έχω την εμπιστοσύνη σας και συγχρόνως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας και τις ερωτήσεις σας σε αυτή την ακρόαση. Uh, thank Σας ευχαριστούμε κύριε υποψήφια επίτροπε. Έχουμε τηρήσει πιστά το χρόνο μας και κάποιες πληροφορίες. Θα δώσω το λόγο στον Συμπρόεδρο Λαβία για να μας ενημερώσει για τα διαδικαστικά, ιδιαίτερα για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ Γέζη. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές, τον προτινόμενο επίτροπο, για τις ερωτήσεις και απαντήσεις και να ενημερώσω τους συντονιστές της Επιτροπής Περιβάλλοντος ότι η συνεδρίασή μας για την αξιολόγηση, την κοινή αξιολόγηση θα γίνει 10 με 11.30 αύριο το πρωί. Ενώ στις 11.30 με 12.30 θα έχουμε την κοινή συνεδρίαση των συντονιστών των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας, ΕΒΚΕΙΤΡΕ για να αποφασίσουμε. Ευχαριστώ και ξαναδίνω το λόγο στον πρόεδρο Μπούζεκ. Τώρα, για τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Ξέρετε οι συντονιστέ πότε θα συνεδριάσουμε για την αξιολόγηση. Το πιο σημαντικό όμω είναι η επόμενή μας ακρόαση. Στη μια μισή αύριο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ε, Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη, του συμπολίτε μας που μας παρακολουθούν απευθείας. Ε, μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους έλαβα μέρος στην ακρόαση και ιδιαίτερα τον υποψήφιο επίτροπο. Καληνύχτα σας.